Έχουμε λοιπόν διάφορες εκθέσεις. Η πρώτη είναι η έκθεση της κυρίας Ροντρίγκε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των εκθέσεων ε, ετήσιας αύξησης και μετά η έκθεση της κυρίας Ριμπέιρο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την πολιτική απασχόληση και κοινωνικές πλευρές στα ετήσια προγράμματα ανάπτυξης, 16 και η έκθεση Στήλε η καθοδήγηση της εσωτερικής αγοράς στα πλαίσια του εξαμήνου 16. Και η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία εισηγήτρια, η Σοφία Ριμπέιγο. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Η έκθεση για τις κοινωνικές πλευρές και την απασχόληση θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια σύγχρονη κοινωνική Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα ε, τι προκλήσει και τι δυνατότητε που έχουμε. Υπογραμμίζει με συγκεκριμένο τρόπο τι πρέπει να εφαρμοστεί για να εξισορροπήσουμε τα οικονομικά με τα κοινωνικά και να υπάρξει ένα κοινωνικό σχέδιο βιώσιμο. Το οικονομικό πιστοτικό σύστημα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ζωή των ε, πολιτών μα. Και αυτό είναι ο κύριο λόγο για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε την ε, εδραίωση αυτών των συστημάτων έχοντας ως στόχο την βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης που πρέπει να περνάει ε, ως κόκκινο νήμα από όλε τις πολιτικές της Ένωσης προτείνουμε να επιτηρούμε την εφαρμογή όλων των πολιτικών από κοινωνική άποψη χρειαζόμαστε όλα τα κράτη-μέλη να εγγυηθούμε με επεύθυνο τρόπο την, ε, των επιλογών μας και στην πολιτική ε, και στα δημοσιονομικά για να έχουμε ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη κατοχυρώνοντα τα δημοσιοοικονομικά και τα φορολογικά μα συστήματα λόγω τη οικονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών που είναι ακόμη πολύ ευαίσθητη πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την εδραίωση για να εγγυθούμε την κοινωνική γαλήνη και σταθερότητα όχι μόνο τώρα αλλά και εν ώψη των μελουσών γενεών. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα να αντισταθούν στην κρίση τα κράτη-μέλη στη, στηρίζεται στη δημοσιονομική τους ε, στεναρότητα. Οι πιο ασθενείς χώρες με τα υψηλότερα ελλείμματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Άρα η δημοσιονομική ε, ε, εδραίωση πρέπει να, να συνοδεύεται και από διαθροτικά μέτρα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εδρεωθεί επίσης ο κοινωνικός ρόλος του κράτους και αυτό είναι πολύ βασικός και, και απειλείται. Η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας και των ε, συνταξιδοτικών ταμείων είναι ίσως το πιο συγκεκριμένο και αυτό παράδειγμα αυτών των προκλήσεων επειδή έχουμε την γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού η οποία θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια και η εκπαίδευση είναι θεμελιώδης τομέας της ε, ανάπτυξης των κοινωνιών μας γιατί έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε στους νέους τις αναγκαίες δεξιότητες για το μέλλον, ιδιαίτερα στους νέους τομείς δραστηριοτήτων, για παράδειγμα στην ψηφιακή οικονομία, την πράσινη οικονομία και την γαλάζια οικονομία. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι όντως ουσιώδεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των επιχειρήσεων, που οι επιχειρήσεις είναι ο κύριος κινητήρας της ανάπτυξης. Επίση, ε, η βελτίωση τη κοινωνική κατάσταση πρέπει να βασιστεί και σε βελτίωση των επενδύσεων και δημοσίων και ιδιωτικών, η οποία πρέπει να στοχεύει προγράμματα που να επιτρέπουν και επιστροφή, δηλαδή ε, το αναγκαίο κέρδος και οικονομικό αλλά και κοινωνικό από τις επενδύσεις. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλώς να διατίθενται δημόσιοι πόροι οι οποίοι μπορεί κατόπιν να στραφούν στην κερδοσκοπία ή στην ε, απόσυρση από την πραγματική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και κοινωνικού δείκτες, για παράδειγμα δείκτη ε, απασχόλησης, δείκτη απασχόληση των νέων, μακροπρόθεσμη απασχόληση, για να μπορούμε να αναλύσουμε συνολικά την κατάσταση των κρατών μελών από κοινωνική άποψη. Αν εγκριθεί αυτή η έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή λέγοντα ότι πέραν των δικτών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών που έχουμε ήδη, χρειαζόμαστε και μηχανισμού που να μα επιτρέπουν να δούμε σε τι βαθμό οι πολιτικέ μα έχουν επιπτώσει στι συνθήκε της καθημερινής ζωής των συμπολιτών μας. Έτσι θα εγγυηθούμε την εσωτερική ισορροπία των κρατών μελών, ούτως ώστε να ε, ε αναπροσανατολίζονται οι οικονομικές και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις αν χρειάζεται. Έτσι θα ενισχύσουμε πιστεύω τον κοινωνικό πυλώνα. Τέλος, τέλος. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους κοιόδης των άλλων πολιτικών ομάδων που ε, ε με πολύ μεγάλο ε, με πολύ μεγάλη δέσμευση σε αυτή τη δικασία καταλήξουμε σε κοινή θέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η πρόεδρο. Και η κυρία Μαρία Ζουάου Ροντρίγκε επίση ε, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διότι σήμερα στο Κοινοβούλιο συζητούμε τρεις σημαντικές εκθέσεις οι οποίες αφορούν την κατάσταση, μια μοναδική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη μία κρίση μετά την άλλη και αν θέλουμε να τι αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις θα πρέπει να ενισχύσουμε το, την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον η ανάκαμψη θα είναι ισχυρή και ισορροπημένη. Έχω την χαρά σήμερα να σας παρουσιάσω την έκθεση η οποία εγκρίθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους μου διότι πιστεύω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν πολύ χρήσιμο συμβιβασμό με πραγματική προστιθέμενη αξία για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφετηρία για την έκθεση είναι ε, η δήλωση ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο πρέπει να αξιοποιηθεί για να συνεχιστούν οι προσπάθειες επαναξισορρόπησης, ισοσκέλησης του προπολογισμού και επίσης η επιδίωξη των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Στόχος επίσης είναι η εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση διότι τελικά το μέλλον της Ευρώπης κατ' εμάς θα εξαρτηθεί ακριβώς από αυτού του είδους την ανταγωνιστικότητα που θα είναι μακρόπνοη, θα βασίζεται στην ενεργειακή μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις και θα δημιουργεί καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αν είναι έτσι τα πράγματα βέβαια, θα πρέπει αυτό το μείγμα πολιτικής να στηρίξει αυτές τις φιλοδοξίες και αυτό σημαίνει ότι στο μείγμα πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν ε, ε, στο προσεχές έτος, η τόνωση των επενδύσεων θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εφιστάμενα εργαλεία, αρχές από το επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά βέβαια σημαίνει και ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ε, για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ε, ΜΜΕ ε, σε δάνεια. Χρειάζονται και οι μεταρρυθμίσεις, θα έλεγα οι μεταρρυθμίσεις δεύτερης γενιάς, δηλαδή πρόθεση καινοτομίας, εκπαίδευσης, χρηστής διακυβέρνησης, βιώσιμων συστημάτων πρόνοιας επίσης και θα πρέπει αυτήν την ισοσκέληση του προπολογισμού να την προωθήσουμε κατά τρόπο ώστε να μην υπονομεύσουμε τις στρατηγικές επενδύσεις και την πρόοδο που θέλουμε να περιμένουμε. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. Και βέβαια υπάρχει και η προσφυγική κρίση. Πιστεύω όμως ότι η μεγαλύτερη αξία της έκθεσης έγκυται στον τρόπο ε, διαχείρισης της Ευρωζώνης. Ε, αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωζώνη είναι μια οικονομική οντότητα, Χρειάζεται λοιπόν και το κατάλληλο μείγμα πολιτικών. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι το επενδυτικό κενό που υπάρχει στην Ευρωζώνη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό μπορεί να γίνει με επιμερισμό των συμμετοχών των διαφόρων χωρών. Ιδίω για όσε χρειάζονται περισσότερο διοσονομικό χώρο, περισσότερα περιθώρια Σίγουρα η μείωση των μακροοικονομικών ισορροπιών είναι σημαντική γιατί οι πιο ανταγωνιστικές χώρες θα πρέπει να διευρύνουν την εσωτερική ζήτηση. Από την άλλη πλευρά όμως οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες από την πλευρά τους πρέπει να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα όχι ε, μειώνοντας τους μισθούς ε, ε, και υποβαθμίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες αλλά επενδύοντας στο μέλλον. Αυτά είναι σημαντικά συμπεράσματα. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό στην Ευρωζώνη να υπάρξει μια σύγκληση προς τα πάνω. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει και δημοσιονομική δυνατότητα και βέβαια εφόσον ολοκληρωθεί και η Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρίτη συγγήτρια η κυρία Κατρίν Στήλερ. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο που παρίσταται εδώ. Βλέπω ότι η πρώην συνάδελφο του Κοινοβουλίου είναι εδώ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Η νέα αγορά είναι πολύτιμος πόρος για την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωση τώρα και στο μέλλον. Υπάρχει δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται στην νέα αγορά. Εκτιμάται στο 1-3 ευρώ σε αξία και είναι μια δυνατότητα και ένα ένα συναγερμός για να ξυπνήσουμε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία αγορά και να ωφεληθούμε. Κρίμα που εξακολουθούμε να μην χρησιμοποιούμε τι ε, προόδου που επετέφθησαν τα τελευταία 20 ετία. Βλέποντας ότι ε, υπάρχει παγκόσμιο ανταγωνισμό και διεθνοποίηση οικονομία. Η ενιαία αγορά έχει πολύ μεγάλο δυναμικό για την ανάπτυξη και τι απασχόληση και αυτή η προοπτική έγινε αποδεκτή ευρέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά επανειλημμένε εκκλήσει όμω για την ενίσχυση τη ενιαία αγορά στο Συμβούλιο, και όσον αφορά τι αιτήσεις εκθέσεις και τις καταχώρασεις τάση, δεν έχει επιτευχθεί επαρκή πρόοδο μέχρι τώρα για να έχουμε αποτελέσματα για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα πρέπει να ολοκληρωθεί περαιτέρω η ενή αγορά και θα συνοδεύεται αυτή η αποκαλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών. Η ενή αγορά θα πρέπει να συμπεριφθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο. Τακτικό διάλογο, συμμορφώσεω με τα κράτη-μέλη, σωστή συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου, μία ε, προσέγγιση σφαιρική που θα καλύπτει όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωζώνη και αυτέ που δεν στην Ευρωζώνη, τα εθνικά κοινοβούλια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί θα πρέπει να συμμετέχουν, είναι κρίσιμο για την ιδιοκτησία του όλου προγράμματο και τη διαφάνεια και για την επιτυχία τη όλη διαδικασία. Πιστεύω επίση ότι η εφαρμογή και η υλοποίηση ήδη ισχύουσα νομοθεσία και από τα 20 κράτη-μέλη ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εκμεταλλευτούμε όλη την ε, δυναμικότητα της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια από του δασμούς, να εφαρμόσουμε σαν την οδηγία περιπηρεσιών, σωστή και έγκαιρη ενσωμάτωση εθνικό δίκαιο και η υλοποίηση των διαφόρων της νομοθεσίας για ε, τις κρατικές προμήθειες, σωστή προσέγγιση για τη δημόσια διοίκηση καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες χρειάζεται. Ήδη παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν εφαρμόζεται σωστά ισχύουσα ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και καθυστερεί ανάπτυξη μια αγορά στην Ευρώπη η αλλαγή δεν θα πρέπει να προέρχεται άνωθεν. Όλοι πρέπει να ενστερνιστούν συμμόρφωση και ενοτροπία τη ενιαίας αγορά. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών. Πολυεπίπεδη ιδιοκτησία θα πρέπει να υποστηρίζεται προπαρική βοήθεια, κατάρτιση και τους αναγκαίους πόρου και ε, πληροφορίε που θα είναι διαθέσιμε σε όλα τα επίπεδα. Ε, προσπάθησα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα καλύψω στην έκθεσή μου και γενικά είμαι ικανοποιημένη με το τελικό κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω τους Σκιώδη για τη συνεισφορά τους. Παρόλο που δεν συμφωνούμε πάντα επί όλων των σημείων, όμως καταφέραμε να πετύχουμε στο τέλος μια συμφωνία. Και πιστεύω και ελπίζω ότι είναι, πιστεύουν και άλλοι συνάδελφοι ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαστε εδώ, σαν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, είναι να εξασφαλίζουμε ότι θα θεσπίζουμε δίκαιου και κατάλληλου νόμου. Από τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Αβώνα έχει μεγαλύτερο λόγο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την θέσπιση νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιρροή μα ότι χρησιμοποιήσουμε εφόσον είμαστε το μόνο ε, δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο, για καλύτερου κανονισμού και καλύτερε αρχέ που θα εφαρμόζουμε. Εκ μέρου τη ομάδα μου ζητώ μικρή αλλαγή στην παράγραφο 46 μέσω τροπολογία, να αλλάξει λίγο διατύπωση. Δηλαδή η αρχή τη καλύτερη ε, ε ρύθμιση και διοίκηση να αναφέρεται στην έκθεση σαν καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια τη διαδικασία και καλύτερη λειτουργία που θα επιτευχθεί έτσι τη ενιαία αγορά και για του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Ελπίζω να με υποστηρίξετε, συνάδελφοι υποστηρίξετε την τροπολογία και το κείμενο στο σύνολό του και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την Επιτροπή Προϋπολογισμών ο κύριος Αχτσουή ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την Προεδρία του Συμβουλίου και τον Επίτροπο. Θα ήθελα να επιμείνω επί του όλου τυπικού και επίσημου χαρακτήρα του εγχειρήματο και δεν έχει πολύ έντονη την ε, κοινοβουλευτική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξάμεινο και λείπει και η φιλοδοξία από την έκθεση των ε, πέντε Προέδρων σχετικά με αυτό. Τούτου λεχθέντος και αναφέρομαι σε αυτά που είπε και η κυρία Ροντρίγκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική είναι ένα συμπλήρωμα, μια προσθήκη εθνικών, ένα άθροισμα εθνικών πολιτικών. Και ο συντονισμός πολύ συχνά παραμένει ε, Και γι' αυτό χρειάζεται να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη που δεν μπορεί παρά να διαβρυνθεί εφόσον οι χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη θα εκφράσουν τη σχετική βούληση. Η Ευρωζώνη χρειάζεται έναν προϋπολογισμό και αυτός ο προϋπολογισμός θα μας επέτρεπε να καταπολεμήσουμε τους ασήμετους κλειδονισμούς και να τις αθμίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται από τα κράτη-μέλη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοδοτική Σταθερότητα επιμερίζει κατά κάποιο τρόπο το υπερβολικό χρέο κάποιων χωρών τη Ευρωζώνη και αυτό που θέλουμε χάρη στον προπολογισμό είναι να έχουμε ένα μείγμα πολιτικών, δημοσιονομική πολιτική να εφαρμόζουμε και νομισματική ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ατουίν. Και τώρα από πλευρά του Συμβουλίου η Υπουργό ε, Ζανίν Χένι Μπλάσετ, ε, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο σε περίοδο κρίσης που έχουμε διάφορα πιεστικά θέματα. Ευχαριστώ που το Κοινοβούλιο βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με το θέμα. Ναι, είναι περίπλοκο. Αλλά πρέπει να μας απασχολήσει με κάθε προσοχή. Γιατί αν θέλουμε η Ευρώπη να σημαίνει κάτι για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, Πρέπει να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για την οικονομική ανάπτυξη και την ε, απασχόληση. Ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίε για του νέου, για του μακροχρόνια ανέργου, για τι μικρέ επιχειρήσει. Και ναι, βεβαίω έχουμε πολλά να κάνουμε. Αλλά η κατάσταση βελτιώνεται. Η Ευρώπη είναι ήδη σε μια αργή αλλά σαφή ανάκαμψη. Βγαίνουμε από την κρίση. Ποιε προτεραιότητε λοιπόν πρέπει να καθοδηγήσουν τη δράση μα σε αυτή τη συγκυρία. Διαβάζοντας τι εκθέσεις σας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με χαρά διαπίστωσα ότι έχουμε κοινή εκτίμηση για τις προκλήσεις ενώπιών μας. Προφανώ. Πρέπει να ενισχύσουμε την ευαίσθητη ανάκαμψη. Και όπως λέει και η συγκίτρια κυρία Ροντρίγιο, το βασικό είναι οι επενδύσεις. Βεβαίως, το σχέδιο επενδύσεων της Κομισιόν είναι κεντρικό στοιχείο της προσπάθειάς μας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, επί του οποίου συνεργάστηκαν Κοινοβούλιο-Συμβούλιο, έχει αρχίσει να λειτουργεί. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Α συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμεθα με την ίδια αίσθηση επίγουσα ανάγκη δράση για να σταματήσουν όλα τα εναπομένοντα εμπόδια και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που να ευνοεί πραγματικά τι επενδύσει. Πρέπει να έχουμε βεβαίω υγιή δημοσιονομικά. Αυτό είναι ουσιώδε στοιχείο τη στρατηγική μα. Γιατί η ανάκαμψη μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο αν βασιστεί σε σταθερό έδαφος. Δηλαδή τα φορολογικά μας πρέπει να ευνοούν περισσότερο την ανάπτυξη και να αναπτύξουμε σύγχρονα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε με ενθουσιασμό τις διαρθρωτικές αλλαγές για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, ούτω ώστε να είναι ανθεκτικές για το μέλλον. Τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα εκείνα που εθίγησαν περισσότερο από την κρίση τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει φιλόδοξες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων που αρχίζουν να δίνουν καρπούς. Ωστόσο, επειδή οι πιέσεις θα αρχίσουν να μειώνονται, μπορεί να επανέλθει ο πειρασμός, ε, να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά επειδή ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα, εάν παραμείνουμε ακίνητοι, θα πέσουμε. Άρα πρέπει να κινούμεθα. Πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τις οικονομίες μας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να διασφαλίσουμε τι αναγκαίε δεξιότητε για του νέου για να αντιμετωπίσουν τι μελλοντικέ προκλήσει. Οι μεταρρυθμίσει λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν την ανταγωνιστική Ευρώπη του αύριο. Στι προσπάθειέ μα να υπάρξει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη πρέπει να βασιστούμε στο ισχυρότερο ατού μα να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε τη ενιαία αγορά. Όπω είπε και η κυρία Στήλα. Ε, είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει διάσταση ενιαίας αγοράς. Βεβαίως, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς είναι κάτι που θέλει να το προωθήσει πάρα πολύ η Ολλανδική Προεδρία και θα κάνουμε μια παρουσίαση γι' αυτό πριν το Συμβούλιο του Μαρτίου. Και βασικό στοιχείο της προσέγγισής μας είναι ότι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση για το αύριο. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες να αντέξουν στις μελλοντικές προκλήσεις. Πώς θα το διασφαλίσουμε αυτό? Πρέπει να επανεξετάζουμε συνέχεια αυτά που κάνουμε. Γιατί μια καλή αρχή δεν αρκεί για να προχωρήσουμε αν δεν εφαρμοστούν όλα όσα έχουμε αποφασίσει. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση του εξαμήνου. Να διασφαλίσουμε ότι όντω θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσει. Και εδώ είναι βασική ευθύνη των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο είναι πολύ ενεργό. Μα πιέζει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Και έχει δίκιο. Ως Προεδρία πιστεύω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει η πίεση μεταξύ κρατών μελών για να αναλυφθούν οι αναγκαίες αλλά ορισμένες φορές οδυνηρές μεταρρυθμίσεις. Περισσότερες πολιτικές συζητήσεις για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την κοινή χρήση των βελτίστων πρακτικών και για να διατηρήσουμε το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό το επόμενο 15 μέρο, πέρα από τις συνήθειες συζητήσεις για τις αιτήσει εκθέσεις προόδου θα κάνουμε συγκεκριμένε συζητήσεις στο Συμβούλιο για την εφαρμογή των αναχώρα συστάσεων φτάνοντας ε, στη συνάντηση κορυφής του Μαρτίου. Όμως, να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει εύκολη λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό στην εφαρμογή. Και δεν θα αρκέσουν περισσότερες και βαθύτερες συζητήσει στο Συμβούλιο. Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατικού ελέγχου είναι ουσιώδες για αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματική. Γιατί το να ενστερνιστούν πραγματικά όλοι αυτοί οι φορείς ε, τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ουσιώδες. Γι' αυτό κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Έχει σημειωθεί λοιπόν πρόοδος. Χρειαζόμαστε όμως ε, πιο επικεντρωμένες συστάσεις για να ασχοληθούμε με τα βασικά θέματα. Και ο ρυθμός ε, του εξαμήνου μας επιτρέπει να επιτύχουμε περισσότερη πολύπλευρη επιτήρηση. Και η έγκριση των συστάσεων για την Ευρωζώνη σημαίνει ότι οι συζητήσει για τι εθνικέ συστάσει από εδώ και μπρο θα λαμβάνουν υπόψη τι προκλήσει που αφορούν ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επίση, ε, θα περισσότερο με την κοινωνική διάσταση του εξαμήνου. Όλα αυτά μαζί είναι ουσιώδει αλλαγέ. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μα για να αποκομίσουμε τα αναγκαία ωφέλη από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με ένα στόχο στο μυαλό μας να υπάρξει ισχυρότερη Ευρώπη για όλους τις, τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα ο Αντιπρόεδρος Βάντης Ντομπρόμσκης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για μια ακόμη φορά. Αξιότιμοι βουλευτέ, σήμερα το πρωί το Σώμα των Επιτρόπων Είχε μια συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, συζητήσαμε και τις εκθέσεις αναχώρα και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Την Παρασκευή ε, θα έχουμε τις εκθέσεις αναχώρα και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Οι εκθέσεις αναχώρα ακολουθούν τις πολιτικές κατευθύνσεις ε, τη ετήσιας επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2016 και τα στοιχεία για την Ευρωζώνη του Πρασινού Νοεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2016 είναι πιο ορθολογικό σε σχέση με το παρελθόν, συμπεριλαμβάνει και την Εθνική Διάσταση και την Ευρωζώνη, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις, στη σύγκληση καθώς και τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαθροτικών Ταμείων και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αποφασίσαμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε φέτος και τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Από έξι περνάμε σε τέσσερις ε, κατηγορίες. Καμία ανισορροπία, ανισορροπία, υπερβολική ανισορροπία και υπερβολική ανισορροπία ε, με διορθωτικό σκέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θέλουμε τώρα να εντάξουμε όλα αυτά στο πλαίσιο του γενικότερου οικονομικού πλαισίου. Υπάρχει ανάκαμψη, αλλά τους τελευταίους μήνες ε, είχαμε κάποιες αρνητικές ε, εξελίξεις στο εξωτερικό. Επηρεάστηκαν ε, οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές, έχει πληγεί κάπως η εμπιστοσύνη Υπάρχει πρόβλημα και με την ανεργία σε πολλές χώρες, ιδίως ό,τι αφορά τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους. Άρα, σε ό,τι αφορά τώρα την προσαρμογή των μακροοικονομικών ανισορροπιών, έχουμε σημειώσει πρόοδο, δεν έχουμε όμως ολοκληρώσει την προσπάθεια, έχουμε ψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους που καθυστερούν πολλές ε, χώρες ε, από το να προχωρήσουν σε ανάπτυξη, αναπτυξιακούς ρυθμούς. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για διπλασιασμό των προσπαθειών για τη στήριξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης και έχουμε πολλά καλά παραδείγματα μεταρρυθμίσεων σε διάφορα κράτη-μέλη. Βλέπουμε όμως ότι εξακολουθεί να μην είναι η ίδια η πρόοδος αναχώρα ή ανατομέα. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει περισσότερη πρόοδος με συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους, εθνικά κοινοβούλια και άλλους εμπλεκομένους φορείς. Και βέβαια σημείο κλειδί είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιοποίηση αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στα κράτη-μέλη. Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα νωρίτερα από ό,τι παλαιότερα, αυτό το στόχο εξυπηρετεί, παρέχει περισσότερο χρόνο για να υπάρχει υπάρξει ένα έντονο διάλογο με τα κράτη-μέλη και του βασικού φορεί, προτού ε, προβούμε εμεί ω Κομισιόν στη δημοσίευση των συστάσεων αναχώρα. Επίση, ο ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει εξελιχθεί. Έχουμε την έκθεση και των πέντε προέδρων για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και την ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2015 για τα βήματα προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη. Είμαι πεπισμένος ότι έχει πρωταρχική σημασία να υπάρξει μια ανταλλαγή ε, κρατικών μέτρων στο πλαίσιο των ε, εκθέσεων αναχώρα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τα πορίσματα των εκθέσεων αναχώρα και η έκβαση της ανάλυσης και ε, των ανταλλαγών που είχαμε αλλά και το πώς προχωρούν τα εθνικά προγράμματα σύγκληση και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα οδηγήσουν ε, και στην τετύπωση των ειδικών συστάσεων αναχώρα για το 2016 που θα εκδώσουμε το Μάιο. Έρχομαι τώρα συγκεκριμένα στις τρεις εκθέσεις που συζητούμε σήμερα και ξεκινώ με την έκθεση Stiller. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να καλωσορίσω τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση ε, με την ε, τις διαρτατικές που χρειάζονται για τη διακυβέρνηση της νέας αγοράς. Αυτές οι μεταθέσεις είναι απαραίτητε σε επίπεδο τομέων επιχειρήσεων για να υπάρξει περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να ε, εμβαθύνουμε στις μεταρρυθμίσεις για να θέσουμε τα θεμέλια για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό μπορεί να το πετύχουμε ε, με μεταρρυθμίσεις αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ε, βελτίωση της εσωτερική αγοράς και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Θέλουμε να μειώσουμε το μεγάλο αριθμό περιορισμών στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στα διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των αγορών αυτών. Είναι σημαντικό κάτι τέτοιο γιατί θα βελτιωθεί ο οικονομικό ιστό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα προσαρμοστούν και θα ε, ολοκληρωθούν, θα ενταχθούν ε, στι ε, αλυσίδε αξία που παγκοσμιοποιούνται όλο και περισσότερο. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην έκθεση της κυρίας Ροντρίγκες, να την ευχαριστήσω και να πω ότι φυσικά και συνάδει με τις απόψεις της Κομισιόν ε, πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ε, καλωσορίζουμε την υποστήριξή σας για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη το 2016 με τις προτεραιότητες που εντοπίζουμε. Επίσης βλέπουμε ότι και το περιεχόμενο και ε, το χρονοδιάγραμμα της υποβολής των συστάσεων έχει βελτιωθεί. Θέλουμε να γίνουν προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο ε, στον τομέα των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να υπάρξει επίση στενό συντονισμό ε, για μια πιο εύρωστη οικονομική ανάκαμψη, για υγιή δημόσια οικονομικά και για αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πρέπει να προωθήσουμε τη σύγκληση με βάση τι καλύτερε δυνατέ επιδόσει στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι ένα από του βασικού στόχου του έργου τη Κομισιόν. Τέλο, Έρχομαι στην έκθεση Ριμπέιρο. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή Ριμπέιρο η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας δείχνει κάποια θετικά σημάδια. Βέβαια, εξακολουθεί να είναι σε υψηλά ποσοστά η ενεργεία σε πολλά κράτη-μέλη, ωστόσο μειώνεται σταδιακά, αυξάνει η απασχόληση στους περισσότερους τομείς και για όλες τις ηλικιακές ομάδες οι νέοι σε μεγαλύτερο ποσοστό ε, μπαίνουν ξανά στην αγορά εργασία, υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει κατάρτιση, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την ανική ανεργία και αποδίδουν καρπού οι προσπάθειέ μα σιγά σιγά. Βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια ε, αποκλήσεων που είχαμε να μειώνονται αυτέ οι αποκλήσει. Ε, λιγότεροι είναι αυτοί που είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. Υπάρχουν κάποιοι κάποιες θετικές εξελίξεις. Επίσης, προώθηση κοινωνικών προτύπων, κοινωνική σύγκληση είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να έχουμε κοινωνική σύγκληση. Δίνουμε περισσότερη σημασία στις κοινωνικές εξελίξεις και στην απασχόληση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουμε την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Τα σχετικά μέτρα, οι δέσμοι μέτρων είναι στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά ε, τον κοινωνικό διάλογο, θέλουμε ε, να ενισχύσουμε το διάλογό μας με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και έχουμε και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, με τις οποίες καλούμε τα κράτη-μέλη να ε, δώσουν λόγο, βήμα και στους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε τους νέους δείκτες απασχόλησης ε, στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση των πολιτικών δημοκρατών μελών. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν συνεχίσει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και είναι εμφανή τα θετικά ε, αποτελέσματα αυξάνουν οι ρυθμοί απασχόληση, Βέβαια θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσει ε, για τη δημιουργία ενό θετικού ε, κλίματο που θα ε, οδηγήσει σε ποιοτικέ θέσει εργασία και περισσότερο στον αριθμό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμοι Βουλευτέ, εδώ ολοκληρώνω την ομιλία μου. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιτροπή περιβάλλοντος ο κύριος Ανδρέη Κόβατσεφ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο στόχους. Την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Αλλά δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τους στόχους όταν οι πολίτες μας δεν έχουν καλή υγεία. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα γι' αυτό. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο όμω θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ούτω ώστε να εφαρμοστούν συστήματα υγείας που ανταποκρίνονται στι ανάγκε των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί μια αξιολόγηση των συστημάτων υγεία, να υπάρχει και ένα εποπτικό σύστημα και να δρομολογηθούν παράγοντες που θα μας βοηθήσουν με να μειώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον της Υπήρου μας. Πιστεύω επίσης ότι η ανασκόπηση της πολιτικής για το 2020 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, διότι η οικολογία και η υγεία μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η κυρία Ίσκρα Μιχάλουδα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, κυρία, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην έκθεσή μας απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, προτείνοντας μέτρα για μια καλύτερη ε, χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Πόρων που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων Ευρώπη του 2020. Η αναθεώρηση του πολιτούς ε, πλαισίου συνδέεται με όλες αυτές τις στοιχείες, όλα αυτά τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Ταμείων, των Διευθυντικών Ταμείων και των πόρων για τις επενδύσεις και πιστεύουμε ότι αυτοί οι πόροι μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους του εξαμήνου και για να συμμορφωθούμε και με τις συστάσεις κατά χώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Πρώτος είναι ο κύριος Μάρκος Φέμπα, ΕΛΚ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αιτήσει εκθέσεις ε, ανάπτυξης ε, της Κομισιόν έχει τρία, τρεις προτεραιότητες επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνη πολιτική στα δημοσιονομικά. Νομίζω ότι είναι καλή αυτή η στόχη όλοι μαζί. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν θα πρέπει να το καταχρώμεθα για να επινοούμε νέους δείκτες που ούτε με την ανταγωνιστικότητα, ούτε με τα σωστά δημοσιονομικά, ούτε με τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν. Και στην ουσία δηλαδή απλώς επιδιώκει να εξοραίσει ορισμένα άσχημα στοιχεία. Δηλαδή, αν δεν μα αρέσουν κάποιοι δείκτες, ε, επινοούμε κάποιου άλλους. Εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί έναντι τέτοιων ε, προσπαθειών. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τους ισχυρού, αλλά να δυναμώσουμε τους αδύναμους. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο, τότε άλλε χώρε επωφελούνται από αυτό. Διότι έχουμε πολύ... Ε, εκτεταμένες ε, εμπορικές σχέσεις. Δεν έχει λοιπόν έννοια να προσπαθήσουμε να μειωθεί αυτό το πλεόνασμα το εμπορικό. Το θέμα είναι και οι άλλοι να αποκτήσουν εμπορικό πλεόνασμα. Και το τρίτον που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε λιγότερους στόχους μέσω των ανακράτος ε, συστάσεων για να μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν. Και ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια που αναφέρθηκε σε πολλά θέματα αλλά παρόλα αυτά μας έδωσε μια ισορροπημένη έκθεση την οποία μπορούμε να υπερψηφίσουμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και πρόεδρος για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Ελίζα Φερρέιρα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Ντομπρόφσκης και κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ομάδα των συναδέλφων που επεξεργάστηκαν το, το, το μέτρο αυτό και την έκθεση αυτή. Σαφές το μήνυμα της εκθέσεως αναφέρει ότι είναι η ώρα να αλλάξουμε το οικονομικό θεματολόγιο της Ευρώπης. Οι παλιές προσεγγίσεις κυρίως όπως γινόταν και στη ΣΥΠΑ μέχρι το 2008 είναι ιστορία. Πρέπει να θυμηθούμε ότι όλες αυτές οι προσεγγίσεις οδήγησαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα συνεργασίας και υψηλά επίπεδα ανεργίας. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες χώρες όπως η Γερμανία έχουν κολλήσει ακόμα στις προσεγγίσεις του 2009. Θα πρέπει να έχουμε κερδοφόρες επιχειρήσεις και αυτό δεν επιτυγχάνεται χωρίς εσωτερική ζήτηση και χωρίς ε, επενδύσεις με χαμηλά επιτόκια. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε βασικά έχει ε, εξαλείψει τη ζήτηση. Αν δείτε πώς λειτουργεί η οικονομία στην Κίνα και στις ΗΠΑ, θα δείτε ότι ε, έχουν κλειδονίσει το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις στρατηγικές επενδύσεις και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, αλλιώς η Ένωση θα χάσει τον έλεγχο της μοίρα της. Η Πορτογαλία είναι καλό παράδειγμα σχετικά με αυτό μπορούμε να συμμορφωθούμε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ακολουθήσουμε πολιτική που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αλλά είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίζουν εναλλακτικέ λύσεις όπως αυτή και να αλλάξουν το βασικό μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε όσον αφορά την νομισματική ένωση μέχρι τώρα. Πρέπει να είμαστε ε, ευφυείς αν θέλουμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα. λένε στα χέρια μας η λύση και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Κυρία Ολρίκε Τρεμπέσιους, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η οικονομική κατάσταση της Ένωσης είναι ακόμη με πολλές ανισότητες ε, συνεχίζεται η κρίση στην ε, Νότια Ευρώπη και αν δεν είχαμε τόσο φτηνό πετρέλαιο δεν θα ήταν δυνατή η ανάκαμψη. Πολλές χώρες έχουν αποσυνδεθεί από την ανάκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμενο από τη μία θα πρέπει να περιέχει ανακράτος συστάσεις και επίσης να προσπαθήσει να επανέλθει η μακροπρόθεσμη ανισορροπία η επιτυχία, δηλαδή η εφαρμογή μέσω των κρατών μελών με συγκεκριμένες πολιτικές ήταν μόνο 25% το 2014. Ανεπαρκής λοιπόν, γιατί είναι θελούσια αυτή η εφαρμογή και βασίζεται στην αρχή της ε, επικουρικότητας. Τα κράτη ε, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους λοιπόν. Αλλά στην Ευρωζώνη η κατάσταση δεν παρουσιάζεται σωστά μέσω διαφόρων τεχνασμάτων ή μέσω διαφόρων στρεβλώσεων του τύπου. Άρα ο στόχος ε, να έχουμε ουσιαστική ισότητα δεν έχει επιτευχθεί. Και στην ουσία η μόνη λύση είναι η εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή ε, υπάρχει η τάση να θέλουμε μια οικονομική διακυβέρνηση για να εφαρμόσουμε την ε, οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν κυδαιμονία από την Ευρώπη. Είναι λάθος δρόμος αυτός. Ευχαριστώ κύριε Τρεμπέσους. Ε, πρέπει να σταματήσετε, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την άλλη, ο κύριος Ραμόν Τρεμόσα Ιμπαλσέλς. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Προεδρεύουσα, κύριε Αντιπρόεδρε, η ομάδα ΑΛΤΕ θεωρεί ότι η έκθεση επιδέχεται βελτίωση και γι' αυτό θα υποβάλουμε για αύριο κάποιε τροπολογίε. Και αν υπερψηφιστούν από το μεγάλο συνασπισμό, ε, μπορεί και να επανεξετάσουμε την απόφαση μα να καταψηφίσουμε. Η εκδοχή της έκθεσης που μιλά για περισσότερη ε, ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες, όπως βλέπετε από το νομικό πλαίσιο, δεν μας ε, ικανοποιεί ιδιαίτερα. Θα επηρεαστούν επίσης ε, τα εμπορικά πλεονάσματα και οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν, θα αντιμετωπίσουν επίσης ε, προβλήματα όσο και οι χώρες που αντιμετωπίζουν ελλείμματα δεν μειώνεται η γραφειοκρατία, δεν εξυγχρονίζονται οι οικονομίε, ούτε έρονται τα εμπόδια ε, για την είσοδο στην αγορά εργασία. Με τι τροπολογίε μα, λοιπόν, προσπαθούμε να κάνουμε πιο ισορροπημένη την έκθεση. Η φορολογική επέκταση δεν αποτελεί πανάκια στη σημερινή κατάσταση. Αναφέρουμε πόσο σημαντικέ είναι οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει, αλλά μόνο εφόσον βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και αν κινητοποιηθούν ιδιωτικέ επενδύσει. Η Κίνα επιβραδύνεται και η ΦΕΔ φοβάται στις ΗΠΑ. Είναι καιρό στα κράτη-μέλη να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. E. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. E. Η κυρία Γκαμπρίλα Τσίμα. Ένα λεπτό. Θέλω να ασχοληθώ με τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα απασχόλησης. Και τονίζω ότι ναι μεν έχουμε ορισμένα θετικά γίνονται δομές, γίνονται συγγνώμη επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια τι σημαίνει επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και όπως και πριν νομίζω ότι η προσέγγιση μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δηλαδή να έχουμε μια σωστή πολιτική για κοινωνική πρόνοια και για απασχόληση δεν εγγυάται όλα αυτά Δηλαδή στην ουσία είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Εάν επανερχόμεθα στη λεγόμενη flexi security, δηλαδή ευελιξία και ασφάλεια, στην ε, ουσία πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η έννοια της flex security είναι ο λόγος που έχουμε τόση επισφάλεια σήμερα στην εργασία. Αν θέλουμε να υπάρξει κοινωνικός πυλώνας, τότε πρέπει να διευκρινίσουμε τι περιεχόμενο θα πρέπει να έχει. Πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές να μην οδηγήσουν σε ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, για τους πρασίνους. Ο κύριος Μπάς Άικχουτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία, για την ετοιμασία της εκθέσεως. Και ευχαριστώ και το σκιώδη εισηγητή που θέλω να ευχαριστήσω. Κύριε Τρεμόζα, με εκπλήσετε κάπως. Λέτε ότι καταψηφίζετε την έκθεση διότι χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία για περισσότερες επενδύσεις. Ακούγατε τους επιφανείς οικονομολόγους του ΟΣΑ που είπαν φέτος ότι χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις η Ευρώπη. Φαίνεται όλο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι και θεσμικά όργανα, οικονομικά όργανα εντό και εκτό Ευρώπη λένε ότι χρειάζονται περισσότερε επενδύσει. Οι φιλελεύθεροι ακολουθούν την παλιά στρατηγική. Λένε δεν πρέπει να επενδύσουμε. Πολύ παράξενη στάση και χαίρομαι που αυτή η έκθεση δίνει περισσότερα περιθώρια για επενδύσει και επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Λέμε επίση ότι η οικονομική θέση της Ευρωζώνης είναι κάτι που να εξεταστεί και η διεθνωτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να ε, έχει στόχο την καλύτερη χρήση των πόρων. Είναι καλές στοιχές αυτές της εκθέσεως που υπερψηφίζουμε και θα ήθελα οι φιλελεύθεροι πραγματικά να αλλάξουν τη στρατηγική τους διότι αλλάζει, προχωράει ο κόσμος. Ah, uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ήχοντ, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Τρεμός Μπαλσάου. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Αγαπητέ συνάδελφε από τους Ολλανδούς Πρασίνους είναι ηρωνία αυτή γιατί στο σχέδιο Juncker 66 φιλελεύθεροι καταψήφισαν και οι Ολλανδοί συνάδελφοι υπερψήφισαν και εδώ το ίδιο θα συμβεί. Ένας από τους βασικούς λόγους που καταψηφίζουμε την έκθεση είναι ο εξής. Θέλαμε να αναφέρεται η λέξη επένδυση Συμφωνούμε ότι χρειάζονται επενδύσεις, αλλά να είναι βιώσιμοι οικονομικά, διότι δεν θέλουμε να πηγαίνει σε αεροδρόμια χωρίς αεροπλάνα επενδύσεις, σε τρένα χωρίς επιβάτες και αυτοκινητοδρόμους χωρίς κυκλοφορία. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε σωστές επενδύσεις και δεν θέλουμε να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να κατασκευάζουν ε, υποδομές φαντάσματα. Διακόπτη πρόεδρος. Αυτό δεν ήταν ερώτηση, λέει πρόεδρο. Σα άφησα να μιλήσετε λίγο παραπάνω. Θα δώσω όμω παρόλα αυτό το λόγο στον κύριο Άικοτ. Κοιτάξτε, πρέπει να επανέλθω στην πρώτη σα παρέμβαση. Είπατε ότι καταψηφίζω διότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι στο ύφο θερότητα στην έκθεση. Και αρνητική διατύπωση για τι χώρε όπω η Γερμανία και η Ολλανδία πλεόνασμα. Αυτό είναι καλό. Και πρέπει να το κάνουμε για τι επενδύσει. Αν μόνο βιώσιμε πρέπει να αναφέρεται και αυτό καταψηφίζεται. Στι διαδοτικέ μεταρρυθμίσει επενδύσει λέμε ότι η βιώσιμη μετάβαση των 100 μελών, των οικονομιών των 100 μελών, πω καλύτερη απόδοση όσον αφορά τι πηγέ, του πόρου, είναι και σήμου σημασία. Αν αυτή είναι η ψηφοφορία ε, κλειδί, αυτό το σημείο μπορείτε να το αλλάξετε το πρόσημο και να το κάνετε συν. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Επόμενο ε, ομιλητή, Μάρκο Βάλι. Δυόμιση λεπτά για το EFDD. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η οικονομική συνταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γεννάται από τις ασφαλμένες προοπτικές και αρχές. Λιτερότητα, πειθαρχία, αυστηρότητα, λιτότητα. Αναφέρεται συνέχεια μεταρρυθμίσεις χωρίς αξιολογήσεις των συνεπειών. Οι περίφημες ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς δημόσια ομοστόνωση παραμένουν κάτι συνεπές. Μία χρεοκοπημένη οικονομική συνταγή χωρίς κοινοτικό νόημα και ακολουθούμε την γερμανική βούληση. Δεν αρκεί να πούμε απλώ όχι στη λιτότητα, πρέπει να είμαι ειλικρινή διανοητικά και να εφαρμόσουμε νομισματικό μέσο, μέσω το οποίο θα υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτέ τι εσφαλμένε πολιτικέ και συνεχώ να ε, συνθλίβουν τα εθνικά συντάγματα. Λοιπόν, χρειάζεται με υψηλό κεφάλι να καταπολεμηθεί η λιτότητα. Θα πρέπει να βασιστούμε στι ε, αρχέ τη της ε, και να τι σώσουμε. Ε, έχουμε την, Βρετανία, την Βρετανία που ε, έρχεται και εδώ να συνα, συναλλαχθεί και να αλλάξει συνθήκε συμμετοχή. Και έχουμε μετά ε, κακέ οικονομικέ πολιτικέ για το ευρώ. Λοιπόν, και θα κυρίσω τι Βρυξέλλε και τη Φραγκφούρτη. Υπάρχουν αδικίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο παραδείγματα πιο συγκεκριμένα των αντιχτύπων των μέτρων. Υπάρχουν αδικίες. Για 20 χρόνια έχουμε ένα νόμισμα ε, που δεν εκφράζει μια πραγματική αξία αλλά ενώνει κάποια κράτη-μέλη με σοβαρές διαφορές οικονομικές κοινωνικές. Λοιπόν, ε, το είχαμε τονίσει αυτό που όταν μπήκαμε. Επί σειρά ετών οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί ε, ε, έχουν χρησιμοποιεί την ισοτιμία που έχει προσαρμοστεί στις οικονομίες της και δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα πλεονάσματα στην, στα ισοζυγιά τους. Δεν κάνει τίποτα ε, σωστό Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ αργά εφαρμόζει ε, τις αρχές για την ε, εξισορρόπηση των διαφορών. Λοιπόν, ήδη αντιμετωπίζουμε σε γεκές χώρες και πρέπει να κάνουν εσωτερικές υποτιμήσεις και δεν μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές για να μειωθούν οι διαφορές. Εδώ και ο Υπουργό Οικονομικό, ο κ. Παντοβάν, το είπε αυτό εδώ και μερικέ εβδομάδε. Δείχνουν, δείχνουν οικονομικέ μελέτε ότι αυτό που λέω ισχύει. Για μία ακόμη φορά του γερμανικού πλεονάσματο δεν αντιμετωπίζεται σωστά στο κείμενο θα ψηφίσουμε. Αντιθέτως, από κάποιες πλευρές νομίζω ότι ε, εξυμνείται. Υπάρχει η ελπίδα της τροπολογίας μας για να ε, στριμώξουμε κάπως την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε κατά πόσο ε, κάποιοι δεν θα αντιμετωπίσουν κατάφασα τις διαφορές που κρύβονται πίσω από αυτήν την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Βάλη. Κύριε Βάλη, σας παρακαλώ, την επόμενη φορά να μιλήσετε λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Στο τέλος ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Για την επόμενη φορά παρακαλώ το έχετε υπόψη σας. Επόμενος ομιλητής, Μπερνάρ Μονό, ENF. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά είναι πλήρως αναποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό το πρόγραμμα θέλει να βάλει σε ζουρλομανδία τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν λειτουργεί αυτό. Ο ΣΑ μειώνει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη και τον πλουθωρισμό. Ενώ είναι τόσο καλές οι προϋποθέσεις, χαμηλά επιτόκια της ε, ε, ΕΚΤ, φθηνό πετρέλαιο, το δολάριο έχει μειωθεί. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξεκινά η οικονομία μας. Πριν από μερικά χρόνια οι φιλευρωπαϊστές, πριν από 25 χρόνια, ε, έλεγαν ότι θα οδηγήσει η Ευρώπη στην πλήρη απασχόληση. Αλλά που έχουμε οδηγηθεί στην ανεργία, στη στασιμότητα, στην λιτότητα, στα κέρδη για τους τραπεζίτες. Δεν λειτουργεί το σύστημα και καλά το καταλαβαίνει Βασίλειο και θέλει να φύγει από αυτή την καταδίκη. Τα ίδια αίτια θα προκαλέσουν τα ίδια αποτελέσματα. Καμία από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνεται δεν θα λειτουργήσει. Στην Ευρωζώνη θα είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό δεν θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Μάλιστα, αυτή ήταν η εκπρόσωπη των ομάδων, λέει η Τώρα περνάμε στους υπόλοιπου ομιλητές. Πρώτος είναι ο κύριος Άνταμ Σέινφελντ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να σχετιστεί και με την αξιολόγηση της διακυβέρνησης της ενίας αγοράς. Δυστυχώς όμως πολλά απομένουν να γίνουν στο πεδίο αυτό. Κυρίες και κύριοι, ζούμε στον 21ο αιώνα που χαρακτηρίζεται από τεράστιες ψηφιακές εξελίξεις, παγκοσμιοποίηση, διεθνής ανταγωνισμός, αλλαγή στην κοινωνική νοτροπία της συμπεριφορά των καταναλωτών. Χαρακτηρίζεται επίσης από την ανάδυση εντελώς νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας που μας ήταν άγνωστες μέχρι τώρα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί στην ενιαία αγορά, αλλά ταυτόχρονα και είναι και πιο σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ως Ευρώπη στις παγκόσμιες αγορές, αυτό που χρειάζεται είναι να ρυθμίσουμε τους όρους ε, της οικονομικής δραστηριότητας, να στηρίξουμε τις νοφείς επιχειρήσεις, ε, να στηρίξουμε την ε, καινοτομία, τις τεχνολογικές βελτιώσεις και εξελίξεις. Θα πρέπει να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης, άρα λιγότερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει επίση να εφαρμόσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη πολύ σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και να καταργήσουμε τους μη δασμολογικούς φραγμούς και οποιαδήποτε προστατευτική πολιτική επίσης να την ακυρώσουμε, να την καταργήσουμε και να εστιάσουμε και στην καλύτερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς που νομίζω είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, τρία λεπτά, Σέρχιο Γκουτιέρρεθ Πριέτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Απασχόληση πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια καλή έκθεση, πολύ καλή έκθεση που ε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Ντομπρόφσκι, τη Επιτροπή, ε, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που εσεί περιγράφετε σε σχέση με το τι βιώνουν οι πολίτε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο χρόνια υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε ανάκαμψη, όπου όμω είναι πολύ βραδία και εντελώ άνηση. Το λένε όλε οι διεθνεί εκθέσει, στον ΩΣΑ για παράδειγμα, και το λέω συνέχεια. Μας λέει όσα ότι από το 10% των πιο πλούσιων ε, μέχρι το 10% των πιο φτωχών η διαφορά έχει εφταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και επομένως ε, ποια είναι η κατάσταση με την οικονομική ε, ανασφάλεια, την κοινωνική ανασφάλεια. Τελείως διαφορετικά πράγματα λέτε. Από τη σοσιαλιστική ομάδα λοιπόν τρία πράγματα ζητάμε κυρίως. Πρώτον, να τονώσετε τις επενδύσεις. Δεύτερον, να διορθώσετε τις υπερβολές ε, της ε, υπερβολικής ε, άκρας λιτότητας. Μιλάμε για διαθωτικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις που πλήττουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Και επίσης ενίσχυση της ευρωζώνης και της κοινωνικής διάστασης, κυρίως του κοινού νομίσματος. Ενίσχυση των επενδύσεων, τόνος των επενδύσεων, αν δεν το καταφέρουμε αυτό, και αν δεν έχουμε μια αντικυκλική πολιτική σε αυτό το κλίμα τη αβεβαιότητα, δεν θα έχουμε διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντο. Έχουμε το σχέδιο ναι. Juncker, που όμω δεν ε, προωθεί αυτέ τι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιτυγχάνει το στόχο. Ξέρετε ότι στη Βρετανία ή στι ΗΠΑ έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια οι επενδύσει, αλλά στην Ευρώπη ε, βλέπουμε μείωση ε, των παγκοσμίων επενδύσεων πέρυσι σε σχέση, παραδείγματο χάρη, με το 2013 ή το 2014. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε Θέλουμε επενδύσεις για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Λίγα ξέρουμε ακόμη για το σχέδιο Juncker, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει ε, τις προσπάθειες των κρατών μελών που έχουν προγραμματίσει αλλά δεν έχουν εκτελέσει πολλές επενδύσεις. Επίσης έχουν υπάρξει υπερβολές στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις και δημιουργούν υποεργασία, πολύ λίγες ώρες ε, ε, εργασιακές συμβάσεις που βασίζονται σε εθελοντικές τελείως διατάξεις και ρήτρες. Επομένως γενικεύουμε και δεν καταπολεμούμε το φαινόμενο αυτό ε, της εργασιακής φτώχειας ε, όπου βλέπουμε πολλοί εργαζόμενοι να ε, πληρώνονται όχι αρκετά για να γεμίσουν το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Και επίσης θα πρέπει να ανακτήσουμε το κοινωνικό μοντέλο. Θέλουμε μια πιο δίκαιη πολιτική, πιο δίκαιη πολιτική αλλά και οικονομικά πιο αποδοτική. Θέλουμε δίκαιες αμοιβέ. Θέλουμε επίσης ε, να πούμε ότι ε, με τις επιδοτήσεις, με τις υποτροφίες και τους σταθεροποιητές θα βοηθήσουμε την κατάσταση. Αν δεν ανακτήσουμε το κοινωνικό μοντέλο, επαναλαμβάνω δεν θα διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Τέλος. Θέλουμε μια καλύτερη ευρωζώνη, ε, μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση. Όπως είπα, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε, ε, διακόπτεται. Μιλάτε Κύριε Κουτιέρεθ, μιλάτε πολύ γρήγορα. Πρέπει να σας διακόψω. Κύριε Κουτιέρεθ, αν συνεχίζετε να μιλάτε τόσο γρήγορα, όσοι δεν ξέρουν Ισπανικά δεν σας καταλαβαίνουν, γιατί οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας ε, μεταφράσουν και επιπλέον υπερεύεται και το χρόνο σας. Την επόμενη φορά λυπάμαι, αλλά θα χρειαστεί να σας διακόψω νωρίτερα. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Στάνισλαβ Όσο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξηγήσετε το θέμα της προσβασιμότητας στις εκθέσεις που συζητούμε στις εθνικές γλώσσες, που δεν έχουμε τις εκθέσεις εθνικές μας γλώσσες. Η έκθεση Ροντρίγκε Φερρυπίν μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, και αυτό δεν είναι καινούριο θέμα, έχω κάποια σχόλια. Και θα ήθελα να εστιαστώ επ' αυτών. Οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Το συζητούμε επί μακρόν το θέμα. Συζητούμε και το δεσμευτικό χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων. Οι συστάσεις είναι δεσμευτικές, διότι εγκρίνονται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και πολύ συχνά εστιάζονται επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Δεύτερον, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί θα πρέπει να αυξήσουμε το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να συντονίσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πολλά κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τις συσταθήσεις μεταρρυθμίσεις, άρα θα πρέπει να εστιαστούμε στο τι πρέπει να γίνει για να πείσουμε τις κυβερνήσεις ούτω ώστε να εφαρμόσουν πράγματι τις συστάσεις αυτές περί μεταρρυθμίσεων. Κυρίως τώρα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη νέα οικονομική χρηματοδοτική κρίση. Η κυρία Ούλα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης, την κυρία Ριμπέρο. Είναι πολύ καλή η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πολύ επικοδομητική για τη σύνταξη της εκθέσεως. Η εξέβρεση συμβιβασμών στο ζήτημα αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Πολλές ανησυχίες ελήφθησαν υπόψη. Πρέπει να πω όμως ότι κατά την άποψή μου η Επιτροπή Απασχόλησης τοποθετήθηκε για την έκθεση περιτησία αναπτύξεως με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αλλάξει, να κοιτάει πιο πολύ προς το μέλλον, να αναγνωρίσει τα επιτεύγματα και να αναφερθεί στα, στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στην αγορά εργασίας για να χρησιμοποιήσουμε το πλήρως δυναμικό που υπάρχει και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη που επανέρχεται με αργό ρυθμό στην Ευρώπη. Βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση η ανεργία μειωνόταν ακόμα το Δεκέμβριο του 2015 κατά 0,1% εν συγκρίση με τον Νοέμβριο του 2015. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή. είναι στο 10,4%, η κατάσταση όμως ε, βελτιώνεται. Το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και να μπουν στο κοινωνικό αποκλεισμό σταθεροποιήθηκε το 2013 και 2014 δεν πρέπει να αγνοούμε την κοινωνική κατάσταση που είναι προβληματική και χρειάζονται πολλές προσπάθειες για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, νέες θέσεις απασχόλησης και έτσι να βρεθεί μια διέξοδος από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Για μένα ήταν αυτό το χτύπημα. Α, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Σας επεσήμανα ότι τελείωσε ο χρόνος αγόρευσής σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο κύριος Βιέγκας έχει το λόγο για ένα λεπτό. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη το 2016 αποτελούν την αφετηρία για μια διαδικασία ε, η οποία δεν μας ικανοποιεί είναι νεοφιλεύθερη προσπάθεια για κυριαρχία στην δημοσιονομική πολιτική των κρατομέλων. Οι κατευθύνσει γραμμέ τη εκθέσεω που πρέπει να ακολουθηθεί από τι κυβερνήσει είναι οι ίδιε παλιέ συνταγέ που μα οδήγησαν στη φτώχεια σε όλη την Ευρώπη και στην ανεργία. Είναι πλήρης αποτυχία να αντιμετωπιστεί η κρίση με δημόσιες επενδύσεις ε, και ε, που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πιο ενεργά στις προσπάθειες αλλά λόγω της μη δημοκρατικής φύσεως της νομισματικής ενώσεως οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η συγκέντρωση του πλούτου επιβάλλονται εις βάρος των εργαζομένων. Μόνο αν απαλλαγούμε από ε, την προσέγγιση αυτή θα έχουμε καλύτερη πολιτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λέει κύριε Λάμπερτ, όπω και άλλοι θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτη τη Επιτροπή Απασχόληση για την ανοιχτή τη προσέγγιση. Εντός διαδικασία πολλοί από εμά ζητούσαμε επιμακρών οι κοινωνικέ διαστάσει, η κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να αναγνωριστούν πλήρω. και ελπίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πραγματική αλλαγή όσον αφορά την οτροπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρέπει να περιμένουμε πολλοί από εμά για να πιστούμε. Οι κοινωνικοί δείκτε είναι πρόσδεκτοι, συμπραγματικοί, αλλά θα έχουν νόημα και πραγματικό αντίκτυπο στην πολιτική. Αυτό θέλουμε να δούμε, θα έχουν αντίκτυπο. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες εντός και μεταξύ χωρών. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι παραπροϊόν της οικονομική δραστηριότητα, αλλά απαιτεί συγκεντρωμένη συγκεκριμένη δράση Καλωσορίζουμε την έκκληση εκθέσεως για επενδύσεις στις υπηρεσίες όπως η υγεία, η περίθαλψη των παιδιών, η στέγαση, η φροντίδα για τα παιδιά και η στέγαση, η κοινωνική δικαιοσύνη θα βοηθηθεί με αξιοπρεπή εισοδήματα και πραγματικά ήρθε η ώρα να καλυφθεί η διαφορά πληρωμής των δύο φύλων και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της φτώχειας. Ελπίζουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος θα επανέλθει με κάθε σοβαρότητα στο διάλογο όταν έχει υποστεί τόσες πολλές βλάβες και ζημίε. Ο κύριος Όφλιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο κάθε χρόνο, τη στιγμή που οι υποστηριχτέ της Ευρωζώνης προβλέπουν ότι έρχονται καλύτερες ημέρες και σύντομα μεγάλη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όλα αυτά που ποτέ τελικά δεν συμβαίνουν. Οι υποστηριχτέ του ευρώ μιλάνε για τη δυνατότητα περαιτέρω διαθετικών μεταρρυθμίσεων και σχεδόν ο καθένα συμφωνεί με τον κύριο Ντράγκη ότι το ευρώ είναι επιτυχία. Βεβαίω είναι πλήρη ανοησίε αυτέ. Η ευρωζώνη με αναπτύχθηκε ε, υπό τις ευνοϊκές συνθήκες του περασμένου έτους. Λοιπόν, από την σύλληψη του ευρώ και τους δείκτες που βασίσαν τις οικονομίες στο 100 το πρώτο τρίμηνο του 1999 έφτασε στα 123 για την Ευρωζώνη 17 χρόνια αργότερα. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου και εμείς είχαμε αλλαγές οικονομίες, φτάσαμε το 137 ε, στην ίδια χρονική περίοδο αυτό το πολιτικό σας νόμισμα δεν λειτουργεί και γι' αυτό πολλοί νέοι δεν έχουν δουλειά. Αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι ότου το ευρώ τελικά το βγάλετε από τον πόνο του, το εκτελέσετε το ΣΥΠΗΝ. Δεχόσαστε γαλάζια κάρτα, κύριε Οφλίν. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να καταλάβω, να μου εξηγήσετε γιατί η λίρα στερλίνα τις τελευταίες ημέρες έπεσε. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε τα νομίσματα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν η ισοτιμία τους. Μετά την ε, κρίση του 2008 μειώθηκε η ισοτιμία και της λίρας και σώσαν περίπου εκατομμύρια θέσεις στη χώρα μας και ενώ χάσατε εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας στην Ευρωζώνη διότι δεν μπορούσαν να κινηθούν το δικό τους νόμισμα οι χώρες. Είναι καλό που μειώθηκε η ισοτιμία της ε, τώρα διότι ε, εξύπνησαν ότι είναι αδύναμο το ευρώ. έχουμε κάποια προσωρινή διόρθωση με, από την πολύ ε, προσωρινή μείωση της αξίας Ελλήνας είναι πρόσδεκτο. Η κυρία το και έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη υποφέρει. Όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο. Μαζική ανεργία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ε, λιτότητα. Θέλετε να υπάρξει περισσότερη ενοποίηση, αλλά το πιστεύετε πραγματικά νομίζω ότι είναι πολιτικέ σκοπιμότητε. Θέλετε να καταργηθούν τα εθνικά κράτη. Παρουσιάζεται την ενιαία αγορά σαν αντίδοτο στη μαζική ανεργία, ενώ κάθε μέρα διαπιστώνουμε το αντίθετο. Κλείνουν επιχειρήσει μετεγκαταστάσει, επισφάλεια για ολόκληρου τομεί τη πραγματική οικονομία. Αυτή η ξεροκέφαλη αυτοικανοποίηση με την οποία ασχολείστε με την ενιαία αγορά, νομίζω δεν ανταποκρίνεται στον απολογισμό πρέπει να τον δείτε τον απολογισμό αυτό με ρεαλιστικό τρόπο. Στην ΙΜΚΟ είπαν απίθανα πράγματα ορισμένοι. Είπαν ότι τα εκατομμύρια μεταναστών είναι ευκαιρία για την Ευρώπη και πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Μα είναι ανεύθυνα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τι επιπτώσει θα έχουν για την αγορά εργασία όλοι αυτοί και στου μισθού. Αναρωτιόμαστε ποιο ωφελείται από το έγκλημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι οικονομίε μα χρειάζονται οξυγόνο, διότι πνίγονται από το συγκεντρωτισμό που επιβάλλει η Κομισιόν και οι εμπειρογνώμονέ τη. Η διακυβέρνηση τη αγορά είναι ξεπερασμένη. Η ομάδα μου είναι κατά. Ο κύριο Κάζα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάρχά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Σοφία Ριμπέιρο, να πω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έδειξε ξεκάθαρα ότι παρήχε στα κράτη-μέλη τα απαραίτητα εργαλεία για να εξέλθουν από την οικονομική κρίση που όμως έχει αφήσει τις πληγές της στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η πρόκληση λοιπόν εντοπίζεται τώρα στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε ότι έχουμε τρεις νέους δείκτες για την απασχόληση στον πίνακα αξιολόγηση στο scoreboard. Για να έχουμε λοιπόν ε, μεγαλύτερη ανάπτυξη και οικονομική και κοινωνική, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες και να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, να δημιουργήσουμε σε όλα τα επίπεδα περισσότερες θέσεις εργασίας. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της μια δέσμη εργαλείων, τη στρατηγική κυρίως ε, την Ευρώπη 2020 και την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Θα πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή και των δύο αυτών εργαλείων εργαλείων να βελτιωθεί και η παρακολούθηση, ο έλεγχο, για να έχουμε ευφυή βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Επίσης πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις ε, πολιτικές ε, αγορά και για τους εργοδότες και για τους ε, αναζητούντες εργασία. Πρέπει να διευκολυνθεί η αναζήτηση εργασία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Γκέπχαρτ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ κύριε Κάζα που σας ακούω που λέτε ότι η ενιαία αγορά είναι βασικός πυλώνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά πάντα εκπλήσωμαι όταν ακούω ότι ξεπερασμένες ιδέες εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένους λένε ότι είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι μόνο να γίνεται business και κυρίως από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όλα θα πάνε μια χαρά. Όχι, όχι. Χρειαζόμαστε μια πολύ πιο ολιστική προσέγγιση. Όπως ε, υπόθηκε, ολιστική. Να μην ασχολούμεθα μόνο με την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αλλά να θέλουμε υψηλού επίπεδου θέση εργασίας, προστασία των καταναλωτών στο υψηλότερο επίπεδο. Μόνο τότε όταν αντιμετωπίσουμε όλα αυτά από κοινού, θα μπορέσει η οικονομία μας να προχωρήσει. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν μόνο θέσεις εργασίας, αλλά να υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη. Το οποίο χρειάζεται η κοινωνία μας. Και χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους στην ε, εσωτερική αγορά και εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πλευρές του θέματος και χαίρομαι πολύ. Θα χαρώ ακόμη περισσότερο αν επιτύχουμε να λύσουμε ένα μικρό πρόβλημα με το άρθρο 46 αλλά να μπορέσουν όλοι να συμφωνήσουν σε μια κοινή προσέγγιση. Ο κύριος Λούκε, 1,5 λεπτό. Ο κύριος Λούκε, ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι τμήμα της απόπειρας να καθοδηγηθεί η οικονομική πολιτική της Ένωσης. Η καθοδήγηση της οικονομίας μπορεί να γίνει, κανείς αν έχει, μπορεί να γίνει αν έχει κανείς αρχικό στόχο. Κάποτε είχαμε στόχο. Είχαμε στόχο σταθερότητα των δημοσιονομικών, την, ε, τον εύρωστο χαρακτήρα των οικονομικών πολιτικών. Όμως δεν τον επιτύχαμε αυτό το στόχο. Αντίθετα, κατέρευσε αυτή η προσπάθεια με την κρίση ε, του δημοσίου χρέους το 2007. Οπότε έχουμε τώρα νέα φιλοσοφία. Βάζουμε και άλλους στόχους. Βάζουμε στον κατάλογο αποτελεσμάτων και άλλους δείκτες. Όπως είπε άνθρωπος Γκέπχαρτ, τι ωραία, είπε ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Αν έχουμε πολλούς στόχους, θεωρείτε ότι θα τους επιτύχουμε. Αυτή η προσπάθεια καθοδήγηση οικονομία δεν έχει καμία ζώνη. Τι συμβαίνει σήμερα, καμία έννοια. Τι, τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρωζώνη. Οι στόχοι αγνοούνται. Η Πορτογαλία, λέμε, πρέπει να κάνει οικονομίε, αλλά οι Πορτογάλοι μόλι ενέκριναν έναν προπολογισμό που δεν προβλέπει εξοικονομίε. Και οι Ιταλοί πρέπει να κάνουν οικονομίε. Αλλά λένε ότι θέλουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και θεωρούν ότι μπορούν να έχουν υψηλότερο επίπεδο ελλείμματο. Οι Γάλλοι αποφασίζουν ε, νόμου που σημαίνει ότι για τρίτη χρονιά δεν θα πετύχουν τους στόχους για το έλλειμμά τους. Η Ελλάδα μας κοροϊδεύει και δεν εγκρίνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Να σταματήσουμε λοιπόν όλα αυτά, αφήσουν, να αφήσουμε τις χώρες να κάνουν ό,τι νομίζουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόγκα, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο και, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επίτευγμα της Ένωσης και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δώσει ευκαιρίες και έχει δημιουργήσει απασχόληση και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Αλλά πολλά ακόμη πρέπει να κάνουμε και πολλές προκλήσεις ενώπιον μας. Η διακυβέρνηση νέα αγορά είναι βασική προτεραιότητα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι θαυμάσιο εργαλείο για να το επιτύχουμε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το ρυθμό που ήδη έχουμε μέσω τη συνεταιριστική οικονομία. Οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν νέους τρόπους του επιχειρήν για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ε, επιτύχουν. Πρέπει να συνεργαστούμε για να υπάρχει αναγνώριση της αρχής για να επιτύχουμε την αρχή της, ε, ε, της αμοιβαίας αναγνώρισης και χρειαζόμαστε και περισσότερη νομοθεσία για την επιτήρηση του τρόπου λειτουργία τη αγορά και για την ασφάλεια των προϊόντων. Και καλό την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίε για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λική Πρόεδρο. Ο κύριος Πιμέντα Λόπεθ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα σύνολο κειμένων που επιδιώκουν την εμβάθυνση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Αλλά αυτό που κάνετε κύριε Επίτροπε είναι ότι επιχειρείτε να μασκαρέψετε τις επιπτώσεις αυτών που έχετε κάνει. Μιλάτε για οικονομική ανάπτυξη και για σύγκληση. Αλλά τα όργανα που χρησιμοποιείτε θίγουν την κυριαρχία των, ετών, των κρατών, δημιουργούν ε, κοινωνικές ανισότητες. Είναι επίθεση κατά των κανόνων, είναι επίθεση κατά της προστασίας των εργαζομένων. Απορρίπτουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την οικονομική του πολιτική. Είμαστε κατά κάθε απόπειρα που θα συνεχίσει την πολιτική λιτότητα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η λιτότητα. Πρέπει να ενισχύσουμε αντίθετα την κυριαρχία των κρατών μελών η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη ε, οικονομική πολιτική θα βασιστεί σε, αξιών, ε, σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Δέχεστε κύριε Πιμέντα μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μέλο. Όχι. Καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Ντυρό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ η Πρόεδρος. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο πίνακας βαθμολογίας της Ένωσης, ε, πίνακας επιδόσεων, ε, θέλει να εγγυηθεί καλές επιδόσεις. Έχουμε την ανταγωνιστικότητα, την ε, ανάπτυξη και μεγάλο διοικητικό άκθος. Έχει άλλον ένα στόχο όμως, τη βιωσιμότητα. Όμως δεν αναφέρεται στην έκθεση ούτε η κυκλική οικονομία, ούτε η διαχείριση και η αποτελεσματική χρήση των πόρων, ενώ αυτό είχε ζητηθεί ρητό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2015. Από την άλλη πλευρά, σε μια έκθεση που στόχο έχει τη διακυβέρνηση της ενέας αγοράς, πώς να ε, εξηγήσουμε την έλλειψη μετά το Dieselgate και το σκάνδαλο της ε, Volkswagen να λείπει οποιαδήποτε ε, μνήμα σε έλεγχο της αγοράς ή μετά το LuxLeaks, να μην γίνεται κανένας λόγος για την κοινωνική φορολογική σύγκληση, για τα ισορροπημένα δημόσια οικονομικά. Στρέφω προ την κυρία ε, Στήλερ. Α, πήγαινα προ τα πίσω, κοίταζα, αλλά έρχεστε μπροστά μου τώρα, μάλιστα. Ήθελα να πω ότι ε, δυστυχώς, παρότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, λόγω αυτών των ελλείψεων θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε την έκθεση. Πρόεδρος, αφού την εντοπίσατε πάλι καλά. Κύριε Ντουραν, κύριος Βάμπ, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως κάθε χρόνο Κατά αυτή τη συζήτηση λέμε πολλά για δημοσιονομικά, για νούμερα, για υποτιθέμενες ανισότητες και επικρίνουμε ένα στον άλλον. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης και τα κράτη της Ευρωζώνης έχουν ε, το καθένα την ευθύνη του, ούτω ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ενιαία αγορά με ενιαίες προδιαγραφές και ενιαίους εφαρμοστικούς νόμους. Και δυστυχώ δεν το κάνουν αυτό πολλές φορές τα κράτη-μέλη. Και είναι κρίμα. Γιατί αν όλα τα κράτη-μέλη έκαναν την προσπάθεια να θεωρήσουν ότι η ενιαία αγορά είναι το βασικό θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τότε θα επιτυγχάναμε όντω αυτή την ευημερία. Να μειωθεί το χάσμα ευημερία και η οικονομία θα αναπτυσσόταν όπως πρέπει. Τα λέω κάθε χρόνο αλλά δυστυχώ ε, δεν ακούγονται αρκετά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να τα ξαναλέω. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σούστερ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αυτό το νέο εξάμεινο έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Είναι θετικό ότι υπάρχουν νέε για την ανάπτυξη μέσω νέων επενδύσεων. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όπω και πριν είναι απαράδεκτα υψηλή ανεργία. Και αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Όμως ε, λυπηρό είναι ότι δεν ε, αποκλίνουμε από αυτήν την βλαβερή πολιτική λιτότητα. Ε, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι ακόμη πολύ σημαντικότερη για πολλά από ό,τι καταπολέμηση τη ανεργία. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την απασχόληση, πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Θέλουμε συνεπή πολιτική ανάπτυξη μέσω σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Και θέλουμε μια φορολογική πολιτική που να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπαλλαγή για να έχουμε την αναγκαία χρηματοδότηση. Πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική ζήτηση μέσω επεκτατικής πολιτικής δάνειοδοτήσεων και χρειαζόμαστε να λάβουμε υπόψη περισσότερο τους κοινωνικούς δείκτες στη συστάση πολιτικής. Πρώτη διόρθωση αναφέρεται τώρα έμεσα στο νέο ευρωπαϊκό εξάμεινο, πρέπει να κάνουμε όμως πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμέσμάκερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα της εκθέσεως. Μου φαίνεται λογικό αυτό που αναφέρει. Δηλαδή ότι οι κανόνες και η γραφειοκρατία της τις μικρομεσαίες πρέπει να μειωθεί. Όταν μιλούμε όμως για την κοινωνική οικονομία φαίνεται ότι χάνουμε το στόχο. Για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναμένουμε ο δημόσιος τομέας να δαπανά περισσότερα αλλά λιγότερα. Και αν δακτυλοδεικτείτε τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν ισολογισμένους προϋπολογισμούς, τότε ε, είναι λάθος η στόχευση. Πρέπει να στοχεύουμε τις χώρες που έχουν αύξηση του ελλείμματός σας. Θα πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες επενδύσεις για να καταπολεμηθεί η ανεργία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης, θα απευθύνω το λόγο σε εσά απευθεία. Οι συνταγές που ακολουθήσαμε στην Ευρώπη ήταν υπεύθυνε για τις αποτυχίες που ε, δημιουργήθηκαν από τη λιτότητα και από την αποτυχία να πετύχουμε και να εφαρμόσουμε σωστή κοινωνική και οικονομική πολιτική και αγνώντας τα προβλήματα των διαφόρων χωρών που δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες. Όμως ακολουθούμε μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Όσο πιο μεγάλα είναι τα κράτη-μέλη, τόσο πιο, πολλά, πιο πολλοί μπορούν να παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα της ευελιξής αγοράς εργασίας, την ιδιωτικοποίηση και την αποδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία δεν έχουν αυτά τα ευέλικτα κριτήρια, δεν εφαρμόζονται σε αυτές. Άρα οι προσεγγίσεις είναι αυθαίρετες. Παρ' όλα αυτά, ο Επίτροπος λέει ότι θέλει να συνεχίσει να ακολουθεί αυτό το δρόμο, διότι εκείνοι που θεωρούνται ε, καλοί ε, τελικά είναι αυτοί που πετυχαίνουν τα χειρότερα αποτελέσματα. Κύριος Θάλμπα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ο συντονισμό ε, των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη είναι κλειδί ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε στην, να εγγυηθούμε τη σύγκληση και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, ε, όπως επίσης και να εγγυηθούμε δημόσια οικονομικά τα οποία θα έχουν εξηγιανθεί. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, διότι ο δρόμος προς ε, την οικονομική ανάκαμψη και κυρίως την παγίωσή της είναι οι μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, αναμφίβολα, αλλά και πρέπει να προωθήσουμε την τόσο αναγκαία οικονομική, η ένωση, αλλά και την πολιτική ένωση. Γιατί τι θα πει μεταρρυθμίσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πει ανάπτυξη η Ισπανία, παρά τα όσα λέει η κυρία Ματίας, ε, είναι μια χώρα υπόδειγμα. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσει. αναπτύσσεται σε τριπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με την ε, υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρυσι δημιουργήσαμε 600.000, νέε 600 συγγνώμη, χιλιάδες Πρόεδρος, η κυρία Μπλίνκε Βιτσιούτε για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα ωφέλη μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας και περισσότερων θέσεων απασχόλησης πρέπει πρώτα να γίνουν αισθητά από τους λαούς μας. Αισθανόμαστε κάποια οικονομική ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, να σε επιστήσω την προσοχή επί ενός μεγάλου προβλήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι η φτώχεια των παιδιών. 27% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτωχά. Γι' αυτό θα ήθελα να εθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι μέλη να δημιουργήσουν μια εγγύηση για τα παιδιά. Ένα φορέα με δικό του προπολογισμό και έτσι κάθε παιδί στην Ευρώπη θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην περίθαλψη της υγείας, παιδεία, στέγαση, διατροφή. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη φτώχεια των γυναικών θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να παράσχουν συγκεκριμένες συστάσεις για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των μισθών, των αμοιβών των ανδρών και γυναικών και των συντάξεων. Τη διαφορά συντάξεων ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Όνερ Λένερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην Ευρώπη λέμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς Ανατολάς, προς ε, προς Βορρά, προς Νότο να κινηθούμε και πάντα η ίδια απάντηση. Όλοι θέλουν και δεν υπάρχει απόκριση απόψεων επ' αυτού, στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον. Το κλειδί της αναπτύξεως βρίσκεται στις Βρυξέλλες ή στα κράτη-μέλη. Εκεί υπάρχει απόκληση απόψεων. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάπτει από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της. Και η επιστροφή στην ανάπτυξη έχει ξεκινήσει. Κάποια κράτη-μέλη πηγαίνουν καλύτερα, άλλα λιγότερο καλά. Κατά την άποψή μου, η έκθεση της κυρίας Ροντρίγκε εμπεριέχει καλά στοιχεία για την ενίσχυση της οικονομικής αναπτύξεως στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις, Πρέπει να αυξηθεί η εθνική ζήτηση αν θέλουμε η οικονομία να ξαναμπεί στη σωστή τροχιά. Αυτά δεν θα πρέπει να αποφασίζονται όμως στις Βρυξέλλες. Όλα τα στοιχεία που άπτονται της αναπτύξεως πραγματικά θα πρέπει να προωθηθούν από το Εθνικά Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματα της πολιτικής λιτότητας συμφωνούμε. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όσοι απευθύνουν έκκληση για αλληλεγγύη πρέπει να σέβονται πρώτα απ' όλα τους κανόνες. Ε, και στην Πορτογαλία η ε, λιτότητα ήταν αναπόφευκτη γιατί οι σοσιαλιστές κυβερνούσαν μέχρι το 2009, καταδικάσανε τη χώρα με τις πολιτικές τους, ε, τη χρέωσαν, χρέωσαν τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό λοιπόν από το να επιλέγουμε να προβαίνουμε σε αλόγιστες δαπάνες ε, μέχρι το 9 ε, που μας οδήγησε σε αυτά τα ε, χρέη, τα ελλείμματα και οδήγησε στα ύψη την ανεργία καταλήξαμε στην ε, παρέμβαση της Τρόικας. Είμαστε τώρα όμως το 2016. Οι σοσιαλιστές, οι ίδιοι ακριβώς που κυβερνούσαν, χάσαν τις εκλογές, επιμένουν τώρα όμως ε, παρουσιάζοντας ε, κάποιους προπολογισμού που προσπαθούν να βολέψουν τα πράγματα και ε, τα ξέρουμε αυτά τις ταινίες, τις έχουμε ξαναδεί αυτές. Ε, δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Ευχαριστώ. Έχει... Κύριε Μέλο, έχετε δύο μπλε κάρτες. Μία από την κυρία Ριμπέγου, παρόλο που, που σήκωσε την κάρτα της μόλις ξεκίνησε η ομιλία σας. Αγαπητή συνάδελφε Μέλο, λέει η κυρία Ριμπέγου. Στη συζήτηση αυτή Μίλησε και η κυρία Ροντρίγκε που είχε φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση και μίλησε υπέρ τη ε, ενίσχυση τη Ευρωζώνη. Και από την άλλη μεριά είχαμε την ομιλία του κομμουνιστή συναδέλφου που είναι απόλυτα ευρωσκεπτικιστής. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά απόψεων. Θα ήθελα να μου πείτε εσεί κύριε Μέλου, συμμερίζεστε την απορία μου ε, για ε, αυτόν τον συνασπισμό που άλλα λέει στην Πορτογαλία και άλλα εδώ ο κύριος μα συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν είναι σύμπτωση. Ε, ζήτησα από τον ε, κομμουνιστή συνάδελφο να μου πει αν θέλει να απαντήσει ερώτησή μου και δεν τη δέχτηκε. Και έφυγε τώρα. Δεν είναι εδώ. Κοιτάξτε, στην ε, Πορτογαλία ένα κόμμα έχασε τις εκλογές χωρίς να εξάγει κανένα δίδαγμα από τα λάθη του παρελθόντος και εξακολουθεί να έχει αυτή τη στάση άρνησης να ασχοληθεί με τα δημοσιονομικά και κάνει υπολογισμού που δεν έχουν έννοια. όσοι όμω κάνουν τέτοιου υπολογισμού, πολύ σύντομα θα διαπιστώσουν ότι θα χτυπήσουν τον τοίχο. Υπάρχει και δεύτερη μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Παρακαλώ, η κυρία Γοντρίγκε. Ε, κύριε Μέλλον, είναι θαυμάσια αυτά που λέτε. Το πώς παρουσιάζετε την κατάσταση. Εξακολουθείτε το κοινοβούλιο εδώ να το κάνετε χώρο για εσωτερικές πολιτικές πορτογαλικές αντιπαραθέσεις. Δεν είμαστε γι' αυτό εδώ. Το θέμα είναι αν μπορεί κανείς να συνδυάσει την δημοσιονομική υπευθυνότητα με την επάνωδο στην ανάπτυξη και την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση του κόμματό σα για χρόνια δεν επέτυχε κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ θα ήθελα να μάθω εάν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση που είναι στην, τώρα στην εξουσία θα μπορέσει να κάνει περισσότερο όπως και εγώ νομίζω. Ο κύριος Μέλλον, κυρία συνάδελφα. Κάποια στιγμή στην ομιλία σας αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη μεταξύ χωρών που είναι σε καλύτερη, μεταξύ χωρών που είναι σε καλή και μεταξύ χωρών που είναι σε κακή οικονομική κατάσταση. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θέλετε να μιλήσετε για την ανάγκη να γίνουν διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως, έγιναν λάθη ε, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά δεν είναι δυνατόν ε, να μην κάνει κάτι και παρούσα κυβέρνηση για να το υπερβεί. Πιστεύω ότι η δική σας ε, ομιλία θα έπρεπε να είναι πιο μετροπαθής. Ναι, αλληλεγγύη, αλλά χρειάζεται και υπευθυνότητα. Και από αυτή την άποψη το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ακόμη πολλά να μάθει. Έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο, λέει η πρόεδρος, αλλά δύο μπλε κάρτες αρκούν και μάλιστα κάθε εξαίρεση. Ο κύριος Σάντ, 1,5 λεπτό. Το πραγματικό πρόβλημα της ε, οικονομική κατάστασης στην Ευρώπη είναι ότι δεν έχουμε επαρκείς επενδύσει και άρα δεν έχουμε ανάπτυξη. Για να διατηρήσουμε την απασχόληση και τι ε, συνθήκε και του κοινωνικού κράτους ε, δεν κάνουμε αρκετά. Άρα οι νέοι θεωρούν ότι έχει αποτύχει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει λοιπόν η κοινωνική συνένεση. Δεν είναι λαϊκιστικό να συμφωνήσουμε με αυτού που τα λένε, γιατί είναι σωστό αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι αν συμφωνεί κανεί με αυτό ή όχι. Το πρόβλημα είναι πώ θα επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη για να υπάρξουν καλέ θέσει εργασία, για να μην φοβούνται οι ηλικιωμένοι για τι συντάξει του. Δεν χρειαζόμαστε περίπλοκα τεχνοκρατικά προβλήματα για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να σκεφτούμε με πρωτότυπο τρόπο. Και όχι να σκεφτόμαστε μόνο πώ θα τηρήσουμε το σύμφωνο σταθερότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του προβλήματο. Επενδύσει, δημόσιε και ιδιωτικέ διότι οι ιδιωτικές επενδύσεις ακολουθούν τις δημόσιες, όχι αντίστροφα. Οι δημόσιες επενδύσεις υστερούν. Το Ταμείο Juncker είναι θετικό, αλλά δεν μπορεί να αρκέσει. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται σε εθνικό επίπεδο, όταν δεν εξαρτώνται από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Αν βρούμε τρόπο να υπάρξουν εθνικά σχέδια δημοσίων επενδύσεων, τότε θα ενθαρρύνουμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά αυτό θα είναι κατά πάσα πιθανότητα παραβίαση του Συμφώνου σταθερότητα. Θα πρέπει να σα απασχολήσει αυτό. Όχι. Γιατί το βασικό είναι να υπάρξουν επαρκείς επενδύσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει κάτι παράδοξο. Μιλούσαμε πριν τη Συμφωνία Κάμερον Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τώρα Μιλάμε για τις ε, χώρες ε, της Ευρωζώνης, ε, τις διαφορές από τις άλλες χώρες. Και περάσαμε τώρα να συζητούμε μια έκθεση που είναι απαρχιωμένη θα έλεγα, γιατί δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι χώρες της Ευρωζώνης φυσικά και θα πρέπει να διαβιβάσουν την εθνική κυριαρχία του σε μεγαλύτερο βαθμό στις Βρυξέλλες, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση αλλά με υπόψη ναι, την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, σίγουρα και αυτά που γίνονται στην Ευρωζώνη μας ε, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Χρειάστηκε και πριν από 15 χρόνια να σωθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε, το αντίθετο είχαμε. Πρόεδρος, έχετε εγγραφεί στη δικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ, θέλετε το λόγο για μπλε κάρτα. Δέχεται ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη υψηλού επίπεδου Και δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε την οικονομική ανάπτυξη αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Θέτω το ερώτημα. Ε, έχει έννοια η Βρετανία να θυσιάσει υψηλού επίπεδου κοινωνικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν είπα ότι ισχύει αυτό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θυσιάζει τα κοινωνικά δικαιώματα. Αντιθέτω, πιστεύω ότι με αυτή τη συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο εγγυάται ακριβώς αυτό στη χώρα αυτή. Και συμφέρει και τη χώρα μου αυτό. Διότι αν δεν υπάρχει ισοτιμία όσον αφορά τι κοινωνικέ παροχές, τότε θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα εις βάρος άλλων χωρών. Αυτό που ο Ντέιβιτ Κάμερον κατάφερε είναι το μεγαλύτερο δώρο για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι σε χώρες όπως η δική μου θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Να εγγυόμεθα τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε αυτή, αυτές οι αρχές δεν θα μπορούσαν τελικά να επιβιώσουν. Για ένα λεπτό, κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για όλη τη βοήθεια που μας δίδει αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη αν δεν μιλήσω για τα μέγιστα συστήματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή που ακόμα και το Συμβούλιο θα πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνες του για την εφαρμογή του πακέτου για την εποπτεία των προϊόντων και όσον αφορά την ασφάλεια ε, του θέματος αυτού. Χρειαζόμαστε μια ασφαλή αγορά, χρειαζόμαστε πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν πράγματι ε, πώς επενδύουν, τι επενδύουν, ε, τι αγοράζουν, ε, τι φοράνε μάλλον, σε τι επενδύουν κλπ. Πρέπει να υπάρχει ανεχνευσιμότητα. Δυστυχώς αυτό το πακέτο έχει μπλοκαριστεί για μία ακόμη φορά. Χρειαζόμαστε το Made in αναφέρεται η προέλευση. Υπερασπίζουμε και το Made in Italy και το Made in Europe. Γι' αυτό θα πρέπει το Συμβούλιο να κάνει μια αλλαγή πορείας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε, διαφορετικά δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο κύριος Ντάντι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Προέδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Η ενιαία αγορά αντιπροσωπεύει αναφυσβήτητα το καλύτερο αποτέλεσμα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αξία της φαίνεται από τη συζήτηση αυτών των ημερών όσον αφορά τον Brexit και αντιπροσωπεύει το πραγματικό επιχείρημα εκείνων που στο Λονδίνο θεωρούν ότι δεν είναι σκόπιμο να φύγει το ΕΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσε μελέτε για το κόστο τη μη Ευρώπη δείχνουν ότι η ενιαία αγορά σήμερα είναι ατελή, αλλά έχει τεράστιο δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται. Αλλά σωρεύονται και άλλα σύννεφα στον ορίζοντα σήμερα συμφέροντα και εθνικοί εγωισμοί και η αμφισβήτηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σέγγεν μπορούν όχι μόνο να θέσουν τροχοπέδι τελικά στην μεγαλύτερη ολοκλήρωση αλλά να υπονομεύσουν και τα επιτευθέντα μέχρι τώρα. Ακριβώς αυτή τη δύσκολη στιγμή για Ευρωπαϊκή Ενότητα θα πρέπει να στραφούμε και να εξετάσουμε την έννοια αγορά, να τον θεωρήσουμε κινητήρα ανάπτυξης και καινοτομίας για μια Ευρώπη που θα είναι εκ νέου ανταγωνιστική. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κραστοντεύσκη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι στην οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει και κοινωνική διάσταση. Αλλά τις κοινωνικές πολιτικές σε ποιο βαθμό μπορούμε να τις ε, συντονίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί απλά να καθοδηγεί. Δεν μπορεί να πάρει από τα κράτη-μέλη τις αρμοδιότητες που έχουν, γιατί η κοινωνική πολιτική είναι εθνική αρμοδιότητα. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να δώσει το 20% ε, για κοινωνικά μέτρα, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ούτε μπορώ να συμφωνήσω με το ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εποπτεύει τις και συμβάσεις στα κράτη-μέλη Πάει πολύ μακριά αυτό. Τα κράτη-μέλη ξέρουν καλύτερα πώ θα λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα. Οι κυβερνήσει αυτέ που πρέπει να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Ευχαριστώ. Σούλτσε, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θεωρήθηκε αντίδραση στην σοβαρή οικονομική κρίση. Οι ανισότητες πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα για να αποφύγουμε νέες κρίσεις. Δύο θέματα είναι σημαντικά. Αυτά τα δύο είναι τα σημαντικά, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, γιατί οι συστάσεις του ήταν λίγες και επιφανειακές και τα κράτη-μέλη δεν τις στήρισαν. Δεύτερον, συζητάμε πολλά τώρα για μια πιο κοινωνική Ευρώπη και για κοινωνικούς δείκτες συχνά αναφέρονται. Στην έκθεση αναφέρονται τρει τέτοιοι κοινωνικοί δείκτε. Η ανεργία των νέων, η μακροχρόνια ανεργία και ποσοστό απασχόληση. Αυτοί οι τρει δείκτε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αλλά επίση καλό να υπάρχουν και άλλοι μακροοικονομικοί δείκτε και να έχουν την ίδια στάθμιση. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ομάδων δικτών. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Η κυρία Γκραπίνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη εισηγήτρια, τους και οδησηγητές και όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν ανθρωπολογίες, Αυτό το έγγραφο δεν είναι τέλειο, αλλά εμπεριέχονται πολλά καλά στοιχεία που οδηγήσουν στη διακυβέρνηση της ενίας αγοράς και την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Αυτή η διακυβέρνηση πρέπει να είναι σωστή, καλή και θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πετυχαίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση, το επίπεδο διαβίωσης κλπ. Χρειαζόμαστε διασυνοριακή ανάπτυξη, πρέπει να τονίσουμε τις θέσεις εργασίας στις φτωχές περιοχές χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα. Έχουμε ε, επίσης και τα Εθνικά Συμβούλια περί ανταγωνιστικότητας που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε όμως μια γενική, μια σφαιρική πολιτική ανταγωνιστικότητας, οι δείκτες είναι σημαντικοί, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, αυτό ήθελα να πω. Χρειαζόμαστε πιο δίκαιο ανταγωνισμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ενισχυθούν. Και αυτή η έκθεση είναι πολύ καλή στον αφορά αυτό. Ο κύριος Ογιαζόφσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι τεράστιος θαυμαστής, μεγάλος θαυμαστής της ευέλικτης χρήσεως του μέσου που συζητούμε. Δεν θέλω να μπω στα πεδία άλλων ε, συναδέλφων. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε κάτι που ίσως δεν είναι στο επίκεντρο της συζητήσεως, άρα είναι κάτι σημαντικό για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και για τη δημοσιονομική ισορροπία. Για τις προσπάθειες που καταβάλουμε επίσης στην Ευρώπη. Είναι οι αμυντικές δαπάνες. Μόνο πέντε χώρες, η Πολωνία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εστονία και η Ελλάδα, μόνο πέντε αυτές χώρες δαπανούν περίπου το 2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Οι άλλες χώρες δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι κάτι που το κόστος αυτός επηρεάζει τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και είναι σημαντικό ποσοστό των δαπανών να το λάβετε υπόψη σας παρακαλώ. Η κυρία Λόπε Φοντάνιε. Συμμερίζομαι τους ε, στόχους κατά προτεραιότητα και τις συγκεκριμένες συστάσεις για την Ευρωζώνη. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι πολίτες μας πέρασαν από πολλές δυσχέρειες και γι' αυτό η εδραίωση της ανάκαμψης πρέπει να έχει αντανάκλαση σε όλη την κοινωνία μέσω περισσότερης απασχόλησης. Για την ανεργία των νέων και επίσης ε, για την μακροπρόθεσμη ανεργία όλα αυτά δημιουργούν κινδύνους ε, κοινωνικού αποκλεισμού και είναι δύσκολο να επανέλθει κανείς στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν τα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευση στις σημερινέ και μελλοντικέ ανάγκες αγοράς εργασία, Με περισσότερη συνεργασία του κόσμου της εκπαίδευση με τον κόσμο της εργασία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ανεργία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο υψηλή ανεργία ενώ έχουμε 2 εκατομμύρια κενέ θέσει εργασία. Δεν είναι δυνατόν 39% των επιχειρήσεων που ψάχνουν για προσωπικό να μην το βρίσκουν γιατί δεν έχει τις ε, κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Ένα λεπτό η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Η ενιαία αγορά δεν είναι μόνο η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το μόνο προσμετρήσιμο όφελος για τα κράτη-μέλη. Σήμερα η ακραία δεξιά και αριστερά αρνούνται την αξία της ενιαίας αγοράς για τα κράτη-μέλη και αυτό δείχνει ότι πρέπει να επεξεργαστούμε την παγίωση της ενιαίας αγοράς σε όλους τους τομείς. Αυτή η αγορά δεν πρέπει να απομονωθεί από τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών. Συχνά αναφερόμαστε στους φορολογικούς παραδείσους και τις επιζήμιες συνέπειες αυτών. Απ' την άλλη πλευρά δεν συζητούμε αρκετά τις κακές πολιτικές που παράγουν τη ζώνη του λικόφωτος όπως το αποκαλώ. Η ζώνη του λικόφωτος δημιουργείται λόγω παράλογης φορολόγησης και μη απαραίτητων κανόνων που πλήττουν τους επιχειρηματίες και περιορίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την απασχολησιμότητα, κάτι που δημιουργεί φτώχεια στις κοινωνίες μας. Δεν έχει νόημα η αγορά αν είναι υπερβολικά αριθμισμένη και η συμμετοχή σε αυτή είναι επαχθής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο κύριος Ροζάτη για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή συζήτηση για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Διότι έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτή τη οικονομική πολιτική στην τελευταία δεκαετία. Από το 2005 στο 2014 το ΑΕΠΑ αυξήθηκε μόνο κατά 7,5% και μόνο 5% στην Ευρωζώνη. Δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη σε τέτοιο βαθμό που κατηγορούνται πολύ συχνά για όλα όσα συμβαίνουν οι Βρυξέλλες. Αλλά είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη ευθύνονται τις περισσότερες φορές για τις οικονομικές επιδόσεις τους. Θέλω λοιπόν να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αυξήσει τις προσπάθειές της και να ασκήσει περισσότερη πίεση στα κράτη-μέλη για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Μιλήσαμε για επενδύσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι επενδύσεις. Η απασχόληση, η τεχνολογική πρόοδος. Άρα στις συστάσεις αναχώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην αγορά εργασίας. Περισσότερο στις, ε, στην απασχόληση, στην τεχνολογική πρόοδο. Διότι διαφορετικά δεν θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνώ στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου, Catch the Πολλά τα αιτήματα, θα δώσω το λόγο σε όσο περισσότερες και περισσότερους μπορώ. Μάλετιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο και την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο χρειάζεται πολύ συντονισμός και αυτό σημαίνει συντονισμός ε, για τις περιφερειακές, τοπικές, εθνικές ε, και ευρωπαϊκές ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει συντονισμός μεταξύ της ε, πολιτικής συνοχής και των συστάσεων ε, προς τα κράτη-μέλη. Να συντονιστούν επίσης οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, να υπάρξουν συνέργειες, να συντονιστούν οι πολιτικές για το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ενέργεια, την αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, τη συνοχή. Αλλά και πρέπει να εφαρμοστούν βέβαια όλες αυτές οι πολιτικές. Ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ιδίως αν ληφθούν υπόψη να τα κράτη-μέλη και τα διάφορα αισθητούτα και ιδρύματα που είναι ε, υπεύθυνα για τις διάφορες πολιτικές αλλά και για τις διαφορετικές οργανώσεις ε, ανάλογα με τη χώρα. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμός. Χωρίς το συντονισμό δεν θα πετύχουμε την εφαρμογή των πολιτικών. Ευχαριστώ. Κυρία Φόρτ δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ κυρία Φόρτ. Άρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές, καθώς η Κομισιόν προτείνει την ίδια γνωστή αποτυχημένη συνταγή. Μερκελική λιτότητα, βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και εφαρμογή του αντικοινωνικού συμφώνου σταθερότητα όμως έτσι δεν πρόκειται να μειωθεί η φτώχεια η ανεργία και η πανάπτυξη που πλήττει τους λαούς του ευρωπαϊκού νότου καθώς και τον ελληνικό λαό. μέσα από το ευρωπαϊκό εξάμεινο η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και η τραπεζοκρατία επεμβαίνουν στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής των κρατών της ένωσης καταργούν τη βούληση των ευρωπαϊκών λαών και εκμηδενίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κοινοβουλίων να διαμορφώνουν ελεύθερα τους εθνικούς προϋπολογισμούς. κυρία πρόεδρε η ελλάδα συνεχίζει να στενάζει κάτω από την πότα της τρόικας που διαλύει το ασφαλιστικό βγάζει στο σφυρί τα σπίτια των ελλήνων κάνει φορομπηχτικό ρεσάλτο στις τσέπες του ελληνικού λαού μειώνει τι συντάξει των απόμαχων της ζωής και διαλύει τους έλληνες αγρότες. αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ κύριε Ντομπρόφσκης, καθώς ο ελληνικός λαός εντείνει τον αγώνα του για να πετάξει την τρόικα επιτέλους έξω από την ελλάδα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πρόβλημα γιατί είναι ανεπαρκή σε πολλά κράτη-μέλη. Τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ιδιαίτερα την πρόκληση που θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί πολλοί προβλέπουν ε, ότι θα επανέλθει η κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θέλει να συνδυάσει μια σειρά από πολιτικές. Αυτό βέβαια δεν είναι απλό Εάν θέλουμε, για παράδειγμα, να υπάρξει προσέγγιση των εκπαιδευτικών ε, προγραμμάτων και να συνδυάσουμε και την κοινωνική περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική ανάπτυξη. Δέχομαι πολλά στοιχεία αυτών των εκθέσεων, αλλά θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ροντρίγκη να δεχθεί τι τροπολογίε τη Άλντε, ούτω ώστε να μπορέσουμε όλοι να την υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριο Σιλικιώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί τη θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού. Και φέτο στι εκθέσει για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο διαβάζω πόσο αυτό βοηθά την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα και πόσο αυτό προωθά την απασχόληση και την ανάπτυξη. Κύριοι συνάδελφοι, απασχόληση και ανάπτυξη δεν είναι η ιστορικά ψηλή αριθμή ανεργία και η κατακόρυφη μείωση του εργατικού δυναμικού στι χώρε με μνημόνια ούτε είναι φτωχοποίηση του πληθυσμού αλλά ούτε και απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και η διάλυση του κοινωνικού κράτους. Στις εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο διαβάζουμε για τα πλεονεκτήματα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης. Ποιου συντονισμού. Παραγνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει μόνο στόχο την πρόθεση των συμφερόντων των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και την πίωση προς τα κάτω των μισών και των κοινωνικών δικαιωμάτων εμεί ω αριστερά απορρίπτουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο γι' αυτό θα καταψηφίσουμε και τις εκθέσει αλλά και την λογική του νεοφιλελευθερισμού της λιτότητα των μνημονίων και τη δημοσιονομική πειθαρχία των λαών. Ευχαριστώ κύριε Σιλικιώτη. Ο κύριος Γοπέ. Ένα λεπτό όπως όλοι. Γοπέ. Mm. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Ροντρίγκε και κυρία Ροντρίγκε μάλλον θέλω να πω λίγα λόγια για το κείμενο που συζητούμε. Πιστεύω ότι εμπεριέχονται κάποια σφάλματα. Είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη να τιμωρούνται λόγω σφαλμάτων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω άμεσο αλυσχετισμό μεταξύ πολιτικής συνοχής και της δημοσιονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Και τα δύο στοιχεία είναι σημαντικότατα, αλλά δεν θα πρέπει με μηχανιστικό τρόπο να λύνουμε αυτά τα προβλήματα όπω θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην θυσιάζουμε ένα στοιχείο υπέρ του άλλου. Είναι θλιβερό που η συγγήτρια δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει αυτή την πτυχή στην γνωμοδότησή τη στο κείμενό της θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι επιζήμια και για την πολιτική συνοχή και δεν θα δημιουργήσει και ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπεράριθμη εισρωή μεταναστών λαθρέων ημί θα έχει βραχυπρόθεσμες δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, ενώ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει την οικονομία λόγω αυξημένης προσφοράς φθηνού εργατικού δυναμικού. κάνετε λάθο αν όχι εγκληματείτε. μέχρι τώρα ένα εκατομμύριο περίπου φθηνά εργατικά χέρια όπω τα ονομάζετε περιμένουν στην ελλάδα να βρουν εργασία στην ευρωπαϊκή ένωση. απατάστε αν νομίζετε ότι βγάζοντα την ελλάδα από τη ζώνη σέγγεν επιβάλλοντα αβάσταχτα μνημόνια και καταδικάζοντά τη σε θάνατο θα σταματήσετε και την αθρώα εισρωή λαθρομεταναστών τζιχαντιστών εγκληματικών ε, ισλαμικών εξτρεμιστών που εκμεταλλεύονται τι προσφυγικέ ροέ για την είσοδό στην ευρώπη όλοι αυτοί αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στι χώρε σα. Πώ θα ανακαλύψετε και θα σταματήσετε έγκαιρα τα εγκληματικά στοιχεία, πώ θα εκπαιδεύσετε, συντηρήσετε, περιθάψετε και εντάξετε τι τοπικέ κοινωνίε τα εκατομμύρια των μεταναστών. Είδε πολλοί από αυτού επιθυμούν να επιβάλλουν δια τη βία το νόμο του Ισλάμ. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, αλλά κοινωνικό, θρησκευτικό, εθνοτικό, πολύ δε περισσότερο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιασλοβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η υψηλή ανεργία των νέων με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Οπότε, δεν λειτουργεί το σύστημα εγγύσεων για τους νέους. Άρα πρέπει να σκεφτούμε νέα μέτρα για να αυξήσουμε την ανεργία των νέων μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που δεν χρειάζεται εγγυήσεις. Επίσης, πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι φτωχοί και πολλές θέσεις εργασίας είναι ιδιαίτερα επισφαλείς και χαμηλά αμοιβόμενες. Βεβαίως ε, χρειάζεται ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να καλύπτεται παρκώς από συστήματα κοινωνικής παρά πρέπει να έχουμε αυτές τις ετήσιες ε, εκθέσεις αναχώρα για να δούμε πώς υπάρχει η ανάπτυξη με βάση αυτούς τους τρεις δείκτες. Αλλά, αλλά να σημειώσω επίσης ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες μπορεί να είναι σωστοί, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εκθέση. Κυρία Κονθάλεφ Πένιας. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα ότι με φωνάξατε. Σα ευχαριστώ, περιπτώσει. Οι προτεραιότητε τη έκθεσης για το εξάμεινο ασχολούνται με ζωτικά θέματα για τα κοινωνικά δικαιώματα και τα εργασιακά. Το κείμενο αυτό είναι απατηλό. Παρουσιάζει τι ίδιε συνταγέ λιτότητας που τόσα χρόνια έχουν κάνει τόση ζημιά στην Νότια Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα άκαμπτη η δημοσιονομική εδραίωση και το, ο στραγγαλισμός των δημοσίων επενδύσεων. Άρα δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρώπη. Οπότε η, το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναδιαπραγματευτεί το σύμφωνο σταθερότητας για να υπάρξει περισσότερη ευελιξία για τις προθεσμίες προσαρμογής για να βοηθήσουμε τις χώρες του Νότου. Έχουμε πολύ υψηλή ανεργία στην Ισπανία και ακόμη και πολλοί εργαζόμενοι είναι φτωχοί και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες ε, τέτοιες ε, περισσότερους τέτοιους δείκτες, περισσότερα υψηλότερα τέτοια ποσοστά. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Τα προβλήματα θα τα λύσουμε εάν βάλουμε στην, ε, ε, στο κέντρο της προσέγγισής μας τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έληξε η διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου και έχετε το λόγο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς κύριε Ντομπρόφσκης. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά την πρόοδο της ε, ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής ή πολιτικών. Σημείωσα δεόντως τα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα από τους ευρωβουλευτές. Η ευρωπαϊκή οικονομία βγήκε από την ύφεση, αλλά ακόμα ε, είναι πολύ μέτρια η ανάκαμψη. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για ανησυχία από ότι πριν από μερικούς μήνες το εξωτερικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί και είδαμε μεγάλη ε, ε, ευμετάβλητο χαρακτήρα της αγοράς των, της χρηματοπιστωτικής. Για να τροφοδοτήσουμε την ανάκαμψη πρέπει να στηρίξουμε την ανάκαμψη με μέτρα και πολιτικές για να προωθήσουμε περαιτέρω ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα στη συζήτηση. Με τα χαράς βλέπω όμως ότι πολλοί από εσά εν γέννη συμμερίζεστε την ολοκληρωμένη μας στρατηγική βάση επενδύσεων, διαθωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνη δημοσιονομικής πολιτικής και φορολογικής πολιτικής. Θέλουμε να βελτιώσουμε το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στην Ευρώπη. Καλωσορίζουμε τη συνσφορά του Ευρωκοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μέσω τακτικών εκθέσεων που υποβάλλονται έγκαιρα, όπως αυτές που συζητούμε σήμερα. Καλωσορίζουμε επίσης την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, στην οποία συμμετείχα την περασμένη εβδομάδα. Σημεριζόμαστε κοινού στόχου, πρόθεση οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόληση στην Ευρώπη και προσβλέπω σε συνεχή καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο σε αυτούς τους τομείς και στο μέλλον. Και σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Χένις Πλασάρτ εκ μέρους του Συμβουλίου έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η εσωτερική αγορά είναι ένα μεγάλο ατού για την ε, παροχή ευημερία, απασχόληση, ανάπτυξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση προ του Ευρωπαίου πολίτε. Η εμβάθυνση λοιπόν τη εσωτερική αγορά είναι προτεραιότητα για την Προεδρία μα. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία και των νέων ε, προτάσεων ε, και τη πλήρου εφαρμογή ε, τη υφιστάμενη νομοθεσία. Ε, πρέπει να πω βέβαια ότι το στάδιο τη υποβολή των προτάσεων ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά διαφέρουν οι απόψει των κρατών μέλων σε σχέση με το πώ μπορεί να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του Ευρώπη στη απασχόληση. Σε πολλά κράτη-μέλη πολλά μάλλον κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι αρμοδιότητα εθνική τα κοινωνικά μέτρα και δεν επιθυμούν να απολέσουν μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Το καλό νέο είναι βέβαια ότι όλα τα κράτη-μέλη τονίζουν ότι θα πρέπει να ανανεωθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να εξακολουθεί να ε, εγγυάται την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ε, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση ε, των ε, επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη ε, τους στόχους ε, της στρατηγικής 2020, καταπολέμηση της φτώχεια, μεγαλύτερη ένταξη αλληλεγγύη. Πολύ τονίσατε τη σημασία της υλοποίηση των συστάσεων αναχώρο. αναχώρα. Με συγχωρείτε. Και φυσικά και δεν μπορώ να, παρά να συμφωνήσω απόλυτα, διότι οι συστάσεις αναχώρα είναι κλειδί για τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Πολλέ φορές δεν είναι κάτι εύκολο, το είπα και στην αρχή. Είναι επώδυνες πολλέ φορές οι μεταρρυθμίσεις, παραδείγματο χάρη στα συνταξιοδοτικά, στην αγορά εργασίας. Ωστόσο δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξαναξεκινήσει η πρόοδος και η ανάπτυξη. Συμφωνώ λοιπόν ότι η εφαρμογή είναι κρίσιμη, είναι σημαντική. Υπάρχουν πολλά σημεία ε, που ακούστηκαν σήμερα, θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας ε, τους επόμενους μήνες. Ε, σύντομα θα υιοθετήσει τις εκθέσεις αναχώρα η Κομισιόν, μελετώντας την κοινωνική κατάσταση, θα μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις, για τις ενδεχόμενες ανισορροπίες. Και εν συνεχεία θα διατυπωθούν οι συστάσεις αναχώρα μέχρι το καλοκαίρι. Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Είναι σημαντική αυτή η φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμενού που κάνουμε τον απολογισμό των πεπραγμένων ε, σε κάθε κράτος μέλος και θέτουμε και τους στόχους για το μέλλον. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν μεταρρύθμιση συστημάτων κοινωνική προστασίας, ε, ρύθμο λειτουργούσε ε, αγορέ, καλέ πολιτικέ για την αντιμετώπιση, παραδείγματο χάρη, της πρόσφατης μαζικής εισόδου μεταναστών και προσφύγων. Για όλα απαιτείται ιδέωσα προσοχή για τα επόμενα χρόνια. Και για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα... στις εισηγήτριες, με πρώτη την κυρία Ροντρίγκες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και ευχαριστώ για τις δηλώσεις ε, της Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τρεις αυτές εκθέσεις δημιουργούν ε, περισσότερη δέσμευση για να υπάρξει ισχυρότερη ανάκαμψη, για να εφαρμοστεί η στρατηγική Ευρώπη 2020 με το σωστό συνδυασμό επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων αλλά για να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες και οι κοινωνικές ανισότητες, κάτι που είναι αναγκαίο. Το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξουν αποτελέσματα στις επόμενες φάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Και γι' αυτό θα πρότεινα ότι με βάση την πολύ θετική πείρα μας των τελευταίων μηνών θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια διοργανική συμφωνία για να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και θα μπορούσαμε σύντομα να έχουμε από τα αποτελέσματα. Μπορούμε να συζητήσουμε κάρποφόρα πριν εγκριθεί και αμέσως μόλις εγκριθεί η ετήσια έκθεση για την ε, ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε με την Κομισιόν Καρποφόρα Κατόπιν είχαμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια που ήταν επίσης μια ευκαιρία για να συζητήσουμε με την Προεδρία του Eurogroup και τώρα εμείς ως Κοινοβούλιο αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να υποβάλουμε τις εκθέσεις μας μάλιστα πολύ έγκαιρα για να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της ε, συνάντησης κορυφής του Μαρτίου του Συμβουλίου. Άρα έχουμε συνεργασία Κοινοβουλίου-Συμβουλίου. Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτές τις προόδους και να κάνουμε περισσότερα. Να εξετάσουμε το δεχόμενο μιας διοργανικής συμφωνίας, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να έχει περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά να έχει και περισσότερη αποτελεσματικότητα για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Χρυμπέιου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το λόγο την, την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πληρέστατη η συζήτησή μας υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, κοινό νήμα που θα πρέπει να ερευνήσουμε, τις επενδύσεις. Η ερώτηση είναι τι είδους επενδύσεις, υπό ποιες συνθήκες θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις. Όλοι φέρουμε ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι κάτι που μέχρι τώρα αποκλειστικά το χειριζόταν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να παράσχουν σταθερότητα στη δημόσια πολιτική. Θα πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όταν μιλάμε για εμπιστοσύνη, αναφέρθηκε εκτενώς η Πορτογαλία, οι συνάδελφοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία για την ψήφο εμπιστοσύνης η οποία έλαβε χώρα και η οποία στήριξε τελικά την κυβέρνηση. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Η κυρία Ροντρίγκε είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και δεν μπορούμε να εξακολουθούμε ε, να συμμορφωνόμαστε με αυτά που απαιτεί η κοινή γνώμη, ούτε να κοιτάμε προς το παρελθόν. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, να εφαρμόζουμε υπεύθυνε πολιτικές να εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν εξεταστεί σωστά. Την τελευταία διετία στην Πορτογαλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομική και η κοινωνική ανάκαμψη έχει ξεκινήσει. Ακόμα σε εμβριακή κατάσταση είναι, αλλά μας δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Όσον αφορά τομείς που πρέπει να επαναξεταστούν, αυτή είναι και ευθύνη μας άλλωστε, για τους τομείς αυτούς πρέπει να του εξετάσουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αυτοσκοπό η αλλαγή. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια, μαζί με του κοινωνικού εταίρου, όλοι μαζί να φτιάξουμε κάτι που θα έχει αποτελέσματα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να δημιουργήσουμε πραγματικά μια Ευρώπη για του πολίτε. Η κυρία Στήλερ. Για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, τους Σκιώδης, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημασία της ενιαίας αγοράς ακούστηκε σήμερα. Και είναι κρίμα να έχουμε ε, μια ενιαία αγορά χωρίς να υπάρχει εξορρόπηση με τα κοινωνικά δικαιώματα. Ισχυρό σημείο της Ευρωπαϊκής Ενώσης Πολύ αναφέρθηκαν στον ψηφιακό τομέα. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό στα τελικά μου σχόλια. Τη σημασία που έχει η ψηφιακή ενιαία αγορά Έχουμε μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε αυτό το τομέα. Δείτε τι γίνεται. Δείτε όλοι έχουμε τα έξυπνα τηλέφωνα. Μέχρι το 2021 71% των τηλεφώνων θα είναι έξυπνα τηλέφωνα, smartphones. Μέχρι το 2020 14 δισεκατομμύρια συσκευές ε, διαδικτύου θα υπάρχουν και αυξήθηκε κατά 65% η κίνηση στην κινητή τηλεφωνία από το τέταρτο τρίμηνο του 2014 με το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Ζούμε μια επανάσταση πραγματική και αυτό συνδέεται με το εξάμεινο και την ενιαία αγορά. Υπάρχουν τρία σημεία που θέλω να θίξω. Το ένα αφορά την προσβασιμότητα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τη σχετική στρατηγική προσβασιμότητα σε πολύ ταχύευρη ζωνική παροχή υπηρεσία. Προσβασιμότητα ούτω ώστε εκείνοι που έχουν όλοι που έχουν και τα ελάχιστα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Δεν θέλουμε αυτό το, αυτή μικρή το ψηφιακό κενό να γίνει ψηφιακό χάσμα. Ε, θέλουμε τελικά να το προωθήσουμε αυτό. Λοιπόν, στην Σκοτία, εκείνοι που θέλουν να δημιουργούν λογισμικό μπορούν να το κάνουν εντός τριμήνου, τετραμήνου. Ε, αυτό αφορά και τη διαβίω εκμάθηση και την οτροπία. Δηλαδή, είτε σε μικρή επιχείρηση, είτε σε πολυεθνική. Όλοι θα πρέπει να γίνουμε ρεαλιστέ όσον αφορά τα ψηφιακά θέματα. Υπάρχει ευκαιρία μέσω του εξαμήνου και τη ενιαία αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η περιοχή στον πλανήτη που έχει τις περισσότερες γνώσεις και είναι η πιο προχωρημένη όσον αφορά τα ψηφιακά θέματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου. Η συζήτηση